Chers collègues, je Αγαπητοί συνάδελφοι, πάρτε θέσει. Άρχεται η συνεδρίαση. Εάν δεν έχετε αντιρρήσει, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Οι αποφάσει ε, των συντονιστών τη 26 Φεβρουαρίου υπάρχουν στο φακέλου φακέλους σας αν δεν έχετε αντιρρήσει. αυτές οι αποφάσεις ε, εγκρίνονται. Θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι κατόπιν ετοιματό σας εστάλει μία πρόσκληση στο Μάριο Σεντένο, τον πρόεδρο του Eurogroup, να έρθει εδώ να συζητήσουμε για τον προπολογισμό της Ευρωζώνης στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το μελλοντικό πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους. Ε, βεβαίως ε, όλοι γνωρίζετε ότι αυτό το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι αναπόσπαστο ε, κομμάτι των ιδίων πόρων. Να θυμίσω επίσης ότι η Επιτροπή Κοντ ε, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής μας στην παρουσίαση τη ειδική έκθεση για τα κοινοτικά ταμεία στρατηγικών επενδύσεων, έτσι ώστε να στεθεί από επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Αυτή η παρουσίαση θα γίνει στις 11 Μαρτίου στο Στρασβούργο στις 8 ε, παρατέταρτο το βράδυ στην Low στην, στην αίθουσα Low n ε, λάβατε τα πρακτικά της 7 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνονται. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Μάνκα που θα παρουσιάσει το σχέδιο έκθεσής του για τις εκτιμήσεις του προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2020. Έχετε το, ρόλο, έχετε το λόγο, συγγνώμη κύριε Σιγητά. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Ε, ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνολικό προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εξαρτάται από την ψήφιση ημί της συνθήκης για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουμε και τη δήλωση της 25ης Δεκεμβρίου του 2018 για την συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου στον κοινωνικό προπολογισμό. Σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί το Brexit, θα πρέπει να προσαρμοστούν όλα τα μέσα, όλοι οι πόροι στον κοινωνικό προπολογισμό. Και θα ήθελα να υποδείξω ένα στοιχείο Κάτι το οποίο συζητάμε τα τελευταία χρόνια. Βρισκόμαστε ενώψη ευρωεκλογών. Και στις Βρυξέλλες έχουμε το παρλαμετάριο μου. Πολλοί προτείνουν να διευρυνθεί σε διάφορες ε, αίθουσες ε, προβολής και έκθεσης ε. εκθεμάτων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνεται λοιπόν εγκαθίδρυση ευρωπαϊκών τέτοιων κέντρων έκθεσης κινητών μονάδων, ώστε ο πολίτης να μην χρειάζεται απαραίτητα να έρχεται στις Βρυξέλλες για να τα δει και να τα θαυμάσει όλα αυτά, να μπορούν αυτές οι κινητές μονάδες να εκθέτουν τα εκθέματα αυτά σε σχολεία, σε διάφορες κοινότητε για να κατανοήσει ο πολίτης καλύτερα πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν θα ήταν θετικό. Θα είχε θετικές επιδράσεις θεωρώ και σε ό,τι αφορά τις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω εν των επόμενων ευρωεκλογών να αναπτύξουμε τέτοιες κινητές μονάδες σε διάφορες ε, χώρες. Τώρα, να κοιτάξουμε τα διάφορα άρθρα σε ό,τι αφορά την κτηριακή πολιτική. Εδώ θέλουμε να υπάρχει μία διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων στο θέμα των ακινήτων. Χρειαζόμαστε να ληφθούν γρήγορα αποφάσεις στο PHS, το κτίριο PHS. Για το κτίριο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους μια απόφαση για το ποιο σενάριο θα ακολουθηθεί και ποια επιλογή θα προτιμήσουμε. Ό,τι και να αποφασίσουμε όμως είναι σημαντικό μέχρι τέλος του χρόνου να εγκαταλείψουν ε, οι υπηρεσίες στο κτίριο αυτό και να μετακομίσουν σε άλλο κτίριο. Και προφανώ γι' αυτό χρειάζονται χρήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα οι πέντε γενικοί διευθυντέ παραβρέθησαν στον Κοινοβούλιο και η κυρία Μίνχου μα εξήγησε τι γίνεται με τις δαπάνες. Στην έκθεση λοιπόν του Γενικού Γραμματέα περιλαμβάνονται και αριθμητικά στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι καθήκον μας στην παρούσα φάση είναι να εξετάσουμε σε βάθος κατά πόσον στέκουν τα αριθμητικά αυτά στοιχεία και να αναζητήσουμε τις βέλτιστες δυνατές λύσεις προκειμένου να διαμορφωθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι δαπάνες και Στη συνέχεια θα συζητήσουμε και με τους κοιόδες εισηγητές ε, το ενδεχόμενο περικοπών. Θα ήθελα τώρα να, να αναφέρω τους τομείς εκείνους όπου ενδεχομένως να μπορούν να γίνουν περικοπές. Καταρχάς, η κτηριακή πολιτική. Η κτηριακή πολιτική εν γέννη, είτε μιλάμε για εξοπλισμό των κτηρίων, είτε μιλάμε για κτίρια καθευτά. Παραδοσιακά στην κτηριακή πολιτική υπάρχει πάντα ένα απόθεμα. Εδώ μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάποιες περικοπές. Το θέμα της επίπλωσης, ε, η κυρία... Η συγκίτρια πρότεινε να γίνουν ε, εδώ περικοπές και θα το προτείνω και εγώ. Επίσης, σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους οδηγού. και εδώ μπορούμε να κάνουμε κάποια εξοικονόμηση πόρων και σε ό,τι αφορά επίσης τα από ταξιδίου των βουλευτών και για τις υπηρεσίες των Συμβασίου Χρονοδηγών. Και εδώ έχουμε σίγουρα αποθεματικό. Ένας άλλος τομέας. Τεχνικές υποδομές. Εδώ μπορούμε να κάνουμε μεγάλες οικονομίες. Ύστερα, στον τομέα των ε, βοηθών των βουλευτών. Σε κάθε θητεία έχουμε ένα αποθεματικό το οποίο δεν εξαντλείται ποτέ. Και αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε ένα περισσευούμενο ποσό. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή να γίνουν κάποιες ε, οικονομίες. Οι γενικοί διευθυντές λοιπόν και διευθύντριες ανέφεραν ήδη που έχουν γίνει οι οικονομίες αλλά και στο Προεδρείο ο κύριος Βίλαν για παράδειγμα επιβεβαίωσε ότι και το Προεδρείο ενδεχομένω να μπορεί να βρει πόρους. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον Γενικό Γραμματέα να εξετάσει το ενδεχόμενο εξέβρεση και άλλων πόρων σε ό,τι αφορά το θέμα της συνεργασίας των θεσμικών οργάνων τώρα, σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά, το εξωτερικό κόστας για τη μετάφραση, τα έξοδα εκπροσωπήσεις, ενέργειας, διοργάνωση συνεδρίων και εδώ μπορούμε να κάνουμε σημαντικές περικοπές. Έχουμε επίσης ε, και τις ε, συνεδριάσεις στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο και στο θέμα των εξόδων ταξιδίου μπορούμε να κάνουμε οικονομίες, ε, για παράδειγμα με τηλεδιασκέψεις, για να αποφύγουμε τα έξοδα ταξιδίου. Μέχρι το έτος 2020 θα έχουμε πολλές μεγάλες επενδύσεις και για πολλέ μεγάλε επενδύσεις μάλλον θα έχουν ολοκληρωθεί πλέον και οι τελευταίε δόσει. Μιλάμε για επενδύσεις οι οποίε ξεκίνησαν το 2016. Θα πρέπει προφανώ και να υπάρξει κάποια συνέχεια. Έχουμε και το έργο IPEX για σύγχρονες τεχνολογίες ασφάλειας στο Κοινοβούλιο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποια ήταν οι δαπάνες από το 2016 για την ασφάλεια των κτηρίων και θα ήθελα να παρακαλέσω την διοίκηση να μας χορηγήσει μια σύνοψη όλων αυτών των εξόδων και δαπανών για θέματα ασφάλειας. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε σε ό,τι αφορά τα προγράμματα για την... τις υπηρεσίες προς τους βουλευτές. Για παράδειγμα, εφαρμογές ενημέρωσης, ε, υποβοηθούμενη εκμάθηση μέσω υπολογιστών κτλ. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε πόσο ακριβώς κόστησαν όλα αυτά τα προγράμματα. Πολλοί συνάδελφοι τώρα γνωρίζουν ότι υπάρχουν βουλευτές, ότι υπάρχουν συγγνώμη, βοηθοί οι οποίοι έχουν δουλέψει για δύο θητείες ε, στο Κοινοβούλιο. Έχουν κλείσει σχεδόν 10 χρόνια δηλαδή προπηρεσία, αλλά του λείπουν μερικέ ημέρε για να συμπληρώσουν τα 10 χρόνια. Και αυτό θα μπορούσε να διακυβεύσει και τι αξιώσει του για σύνταξη. Έχουμε λοιπόν βοηθού που θα συνεχίσουν μετά τι επόμενε εκλογέ. Κάποιοι, ωστόσο, θα εγκαταλείψουν το κοινοβούλιο. Και δεν θα έχουν κλείσει τη δεκαετία που του χρειάζεται και αυτό ενδεχομένω να του προκαλέσει προβλήματα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους, τα Στις 10 Δεκεμβρίου του 2018 έγινε μια συνεδρίαση του Προεδρείου για το θέμα των ασκούμενων και θα ήθελα και εδώ να ζητήσω για μια σύνοψη να μου χορηγηθεί. Αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή από 2 Ιουλίου 2019 προκειμένου οι ασκούμενοι να αμείβονται σωστά όταν δουλεύουν για έναν βουλευτή. Να αμείβονται επαρκώ για να μπορούν να βγάλουν πέρα. Έχουμε και άλλους τομείς ε, όπου οι δαπάνες δεν είναι αποτελεσματικές. Για παράδειγμα, οι προφορικές ε, δηλώσεις ε, διαλογής ψήφου τις οποίε τι μεταφράζουν οι διερμηνείς, αλλά ουσιαστικά ένα στόχο έχουν, να μπορέσει να τα παρουσιάσει αυτά ο κάθε βουλευτή στην εκλογική του περιφέρεια. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω να γίνει μια λεπτομερής ανάλυση αυτών των αιτιολογήσεων ψήφου. Πόσο κοστίζουν τελικά. Και θα συμβούλευα διάφορους άλλους βουλευτές, ε. αν θέλουν πραγματικά να επεξηγήσουν την ε, ψήφο τους, να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα οι γραπτές ε, επεξηγήσεις ψήφου. Δεν χρειάζεται να γίνονται όλα αυτά ε, προφορικά. Έχουμε και το θέμα του εθελούσιου συντεξιδοτικού ταμείου το 2024. Το ταμείο αυτό ενδεχομένω να έχει αδειάσει ήδη, να έχει μείνει χωρί πόρου. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω το ελεκτικό συνέδριο και τους ελεγκτές να ελέγξουν πραγματικά τι γίνεται με το Ταμείο Συνταξιοδότηση. Θα ήθελα να ζητήσω και από αυτούς μια σχετική έκθεση προφανώς. Ένα άλλο στοιχείο. Η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργανών θα πρέπει να είναι απρόσκοπτη. Εδώ έχουμε δυστυχώς κενά. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας. Οι υπηρεσίες ε, οδηγών, διερμηνή ε, μεταφράσει Ο κ. Βίλαντ, για παράδειγμα, ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια ενιαία μονάδα υπηρεσία ασφάλεια για όλα τα θεσμικά όργανα. Εδώ λοιπόν θα μπορούσαμε να δούμε πώ θα μπορούσαμε να οργανωθούμε και να προβούμε ενδεχομένω και σε οικονομίε. Θα παρακαλούσα λοιπόν το Γενικό Γραμματέα να εξετάσει την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, να αναζητήσει περαιτέρω δυνατότητες συνεργασίας. Στο παρελθόν ε, κάναμε οικονομίες ε, της τάξης των εκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διερμηνίας. Δεν έγιναν αντίστοιχα προσπάθειες από τα άλλα όργανα. Εμείς όμως κάναμε ε, προσπάθειες οικονομίας και αυτό το διδάξαμε σε ένα ενιαίο πακέτο για όλα τα θεσμικά όργανα. Ένα άλλο στοιχείο. Χθες ε, συνεδρίασε η Επιτροπή καταπολέμησης ε, σεξουαλικής παρενόχλησης. Εδώ έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ δύσκολες και περίπλοκες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, επί τετραετίας ε, υπήρχε περίπτωση παρενόχλησης ενός ατόμου ψυχολογικής ε, ταπείνωσης. Αυτό μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο. Θα πρέπει λοιπόν να παρατηρήσουμε τα φαινόμενα αυτά και να παρα... παρεμβαίνουμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, πέρσι ορίσαμε έξι αρμόδια άτομα. Μετά τις εκλογές, ωστόσο, θα είναι νέοι ε, οι ευρωβουλευτές, καινούργιοι βοηθοί, καινούργιοι ασκούμενοι. Είναι σημαντικό, λοιπόν, εάν συμβεί κάτι τέτοιο εκ νέου, να υπάρχουν δυνατότητες να στραφεί κανείς στον αρμόδιο, να στραφεί στον διαμεσολαβητή, για να καταγγείλει πάρα αυτά το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί κατευθείαν, να μην υπάρχει αναβολή και προφανώς και προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχοι πόροι. Τα προβλήματα λοιπόν αυτά από εδώ και πέρα θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με επαγγελματικό τρόπο. Ένα επιπλέον στοιχείο τώρα το οποίο αναφέρω και στην έκθεση και το ανέφερα ήδη είναι ότι χρειαζόμαστε πιο πολλέ τηλεδιασκέψει για να αποφεύγουμε τα έξοδα ταξιδίου. Αυτό προφανώ είναι προ όφελο και του περιβάλλοντο και προφανώ και μπορούμε να μειώσουμε τα έξοδα ταξιδίου, γιατί έχουμε και τρει έδρε στο Κοινοβούλιο. Πολλοί συνάδελφοι θα θυμούνται ότι όλη η διαδικασία προπολογισμού θέλαμε να απλοποιηθεί και έχουμε εδώ τα έγγραφα τα οποία τα εξετάσαμε, τα καταρτήσαμε για την διαδικασία απλούσταυση αυτής. Θα ήθελα λοιπόν να δηλώσω το εξή. Μετά την ολοκλήρωση της προεκλογική εκστρατεία. θα ήθελα να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα εργασία η οποία και να συνεχίσει να εξετάζει δυνατότητε περικοπή ε, των εξόδων σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες διερμηνίας, σε ό,τι αφορά ε, τη διοργάνωση του συνεδρίου. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα αυτό το μόντου operandi, αυτό το έγγραφο να το υποβάλω για την διαδικασία καθορισμού του προπολογισμού, προκειμένου όλα αυτά να τα λάβει υπόψη και η επόμενη γενιά, αν θέλετε, η οποία θα προκύψει μετά τις ευρωεκλογέ και να συνεχίσει στα βήματά μα. Μπορούμε λοιπόν να γλιτώσουμε μεγάλα έξοδα και σε ό,τι αφορά τη μετάφραση, γιατί πολλές μεταφράσεις γίνονται περιτά, και σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να παρικόπουν περαιτέρω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ ε, που θα γίνει η συζήτηση και είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι είμαστε σε θέση να υποβάλουμε ένα καλό προπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και αν δεν έχουμε τόσο πολλά μέσα στη διάθεσή μα όπω παλιότερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Σας ευχαριστώ για αυτό το ενθαρρυντικό μήνυμα. εντοπίσατε μια σειρά από ε, ενδεχόμενες ε, δυνατότητες εξοικονόμησης ε, και το Κοινοβούλιο σίγουρα θα βασιστεί στην, παραδειγματικ στην παραδειγματικότητα της διαχείρισης που το ίδιο κάνει. Θα δώσω τώρα το λόγο στους και συγητές. Ο κύριος Ρούμπιγκ έχει αφήσει τον κύριο Φερνάνδη στη θέση του, όχι. Ο κύριος Κιόλμελ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερα τον εισηγητή. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ περιεκτική αυτή η έκθεση, πολύ λεπτομερής και πιστεύω ότι έδειξε και τα πιο σημαντικά στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν. Προσπαθούμε κάπως να τραγωνίσουμε τον κύκλο σε τελική ανάλυση. Συμφωνώ απόλυτα μαζί του όταν λέει ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε πόρους και δαπάνες, κυρίως ε, επικεντρωνόμενοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πιο ουσιαστικά και θεμελιώδη στοιχεία. Έχω επίσης την εντύπωση ότι διάφορες συνεδριάσεις ε, δεν θα ήταν πάντα υποχρεωτικό να διοργανώνονται ή τουλάχιστον ε, με πλήρη με πλήρεις ε, προδιαγραφές. Τουλάχιστον ε, εφόσον δεν έρχονται οι βουλευτές ή δεν έρχονται, εν πάση περιπτώσει, όλοι όσοι υποτίθεται θα έρχονται, θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε πολλά έξοδα μετάφρασης διερμηνίας ε, παράλληλα. Αυτό προφανώ από εμά εξαρτάται. Αν υπήρχε μεγάλη επιταρχία, μεγαλύτερη επιταρχία, θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την έκφραση των στοιχείων αυτών και στα επίσημα έγγραφα. Και επίση το πόσο εκφραζόμαστε. Θα μπορούσαμε να εκφραζόμαστε με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό θα σήμερα μεγάλη εξοικονόμηση εξόδων. Κατά τα άλλα, υπάρχουν ε, και λόγοι για τους οποίους μπορούμε να βγούμε και να υποστηρίξουμε το γεγονός ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούμε να είμαστε και το απάβγασμα της οικονομίας. Έχουμε πολλές υποχρεώσεις, έχουμε τόσα πολλά, τόσους πολλούς επισκέπτες για παράδειγμα κάθε χρόνο. Έχουμε ανάγκη σε προσωπικό και ένα από τα πιο σημαντικά θέματα θεωρώ είναι και το θέμα τη ασφάλεια. Η ασφάλεια στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο συγκεκριμένα. Θα ήταν καταστροφικό πραγματικά αν δεν ακολουθούσαμε το πνεύμα τη εποχή και τελικά ε, βρισκόμασταν αντικείμενα επίθεση. Αυτό πραγματικά θα ήταν πολύ κακό σημάδι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, σε τελική ανάλυση, πιστεύω ότι και οι δυνατότητε εξοικονόμηση είναι σε τελικό βαθμό περιορισμένε. Παρ' όλα αυτά, θα κάνουμε την προσπάθεια που μα αναλογεί. Ευχαριστώ. Sí. Madame Ευχαριστώ, κυρία Γιατεν Μάκη. Έχει δώσει το μήνυμά στον κύριο Ντεπρέ θα την εκπροσωπήσει. Ναι, ναι πρόεδρε και με την ευκαιρία να στήσω συγγνώμη εκ μέρους της ε, είχε άλλες υποχρεώσεις ε, σήμερα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο τον κύριο Μάνκα για το έργο του. Σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα ε, μπόρεσε να κάνει τη δουλειά του. Συμφωνούμε με πολλά από αυτά που είπε, οπότε δεν θα τα επαναλάβω. Ε, θα βασιστώ κυρίως σε κάποια σημαντικά στοιχεία, με βάση και το σχέδιο κειμένου. Θεωρούμε πρώτα απ' όλα ότι ό,τι αφορά τις μειώσεις, τις περικοπές, ο κ. Μάνκα κάποια, Μάνκα κάποια στιγμή είπε ότι θα πρέπει να γίνουν ε, περικοπές σε σχέση με τις προτάσεις του Γενικού Γραμματέα. Η ομάδα μου θεωρεί ότι το συνολικό ποσό αυτών των εξοικονομήσεων πρέπει να ποσοτικοποιηθεί. Προτείνουμε παραδείγματος χάρη το συνολικό ποσό του προπολογισμού για το 2020 να μην μπορεί να αυξηθεί περισσότερο από το δεύτερο του 2019 ε, σε σχέση με το 2018. Το συνολικό ποσό που προτείνεται αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικό. Εάν θέλουμε λοιπόν μια, ένα ποσοστό αύξηση του προπολογισμού του 2020 που να μην είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό αύξηση του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να μπορέσουμε να οικονομήσουμε κάπου 22 με 23 εκατομμύρια. Ε, να το πούμε αυτό. Δεν αρκεί να συμφωνούμε επί της αρχής, πρέπει να διευκρινίσουμε και για ποια ποσά μιλάμε σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση. Άκουσα τον κύριο Μάνκα προηγουμένως ε, ε, να επιχειρηματολογεί υπέρ αυτών των κέντρων ε, ευρωπαϊκής εμπειρίας. Ε, εμείς δεν είμαστε και τόσο ενθουσιώδεις απέναντι στην πρωτοβουλία και θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε να υπάρχει κάποιο κοινοβούλιο σε κάποια χώρα μοσπονδιακή που να έχει κέντρα εμπειρίας ε, στα διάφορα ομόσπονδα κρατήδια. Δεν γνωρίζω τέτοια περίπτωση. Ε, και μου κάνει εντύπωση τώρα, μου φαίνεται περίεργο δηλαδή, ένα κοινοβούλιο, ενώ εκπροσωπεί όλους τους πολίτες της Ένωσης, να θέλει να έχει θηγατρικές κατά κάποιο τρόπο ως κοινοβούλιο, ευρωπαϊκά κέντρα. Εάν όλα τα θεσμικά όργανα τα ευρωπαϊκά, το Συμβούλιο, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο καθόριζαν, ε, έπρεπε να καθορίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρώτα που έχει σημειωθεί, εντάξει, αλλά να υπάρχουν τώρα θηγατρικές έκθεσεις ε, που θα εκτίθεται το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις χώρες, ε, εμεί δεν καταλαβαίνουμε και τόσο ποιο είναι το νόημα αυτής της πρωτοβουλίας και δεν μας ενθουσιάζει. Το λέει και η έκθεση της γραμματείας ότι υπάρχουν μια σειρά από διπλωματικές, ε, διπλωματικά πόστα σε διάφορες χώρες, ε, ε, Τζακάρτα και κάπου αλλού. Ο υπεύθυνο για τη Washington θα είναι επικεφαλής στην Τζακάρτα, κάτι τέτοιο προβλέπεται. Πώς αιτιολογούνται όμως αυτά. Ποια συζήτηση έγινε που οδήγησε στο αποτέλεσμα αυτό και για ποιον λόγο. Εμείς δεν έχουμε κάποια αντίρρηση, αλλά υπάρχουν ήδη πρεσβείες όλων των χωρών της Ένωσης. Υπάρχει υπηρεσία εξωτερική δράσης. Και εμείς ως κοινοβούλιο θα δημιουργήσουμε εκεί καινούργια γραφεία. Ε, είναι αρκετά περίεργο, έτσι. Ε, ορισμένες φορές πρέπει να ρωτηθούμε ε, ποια είναι η σκοπιμότητα κάποιων από τι επιλογέ μα. Να εκπροσωπείται η Ευρωπαϊκή Ένωση από τρία-τέσσερα διαφορετικά διαφορετικές οργανώσεις σε μία χώρα δυσκολεύομαι να το καταλάβω καταλαβαίνετε ενώ είμαι βεβαίως πεπισμένος φεντεραλιστής Ευρωπαίος έχουμε και εμείς κάποιες προτάσεις, προτάσεις εξοικονόμησης ο κ. Μάνκα αναφέρθηκε σε Κάποιου τομεί. Ε, στην προετοιμασία λοιπόν της, της κατάλογου ψηφοφορία θα τα πούμε αυτά. Θα θέλαμε να θυμίσουμε στα πλαίσια τη έκθεση του προπολογισμού του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μια εξυγίανση, του είπε ο Μάνκα, για τη χρηματοδότηση των κτηρίων. Υπάρχει αυτή, αυτή η, η πρακτική τρέχουσα, η οποία είναι νοσηρή. Ε, θα πρέπει να, να δούμε τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση των κτηρίων, διότι υπερεκτιμούνται ε, οι δημοσιονομικέ γραμμές ε, για να μπορέσουμε και να καλύψουμε το κόστος της ενοικίας των κτηρίων. Ε, ε αυτή η πρακτική όμως ε, είναι πραγματικά ανυπόφορη. Κάποια στιγμή ε, θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και αυτό. Να λοιπόν κάποια στοιχεία όπου θα πρέπει να ξεκινήσει μια συζήτηση με τον εισηγητή να δούμε αν θα βρούμε κάποια σημεία σύγκληση. Ε, θέλω να του συγχαρώ για δύο σημεία επίσης. Ε, είναι πραγματικά σκανδαλώδες ε, το ζήτημα αυτών των ε, βοηθών που επειδή τους λείπουν ένα ή δύο μήνε για γραφειοκρατικού λόγους, κάποιοι δηλαδή που δεν μπορούσαν να του ανανεώσουν τη θητεία έγκαιρα, να χάσουν το δικαίωμα τους εξωτικό του δικαιώματα επειδή λείπει ένα μήνα Μετά από δέκα χρόνια Εργασία. σε ποια κοινωνία, σε ποιο κοινωνικό σύστημα ασφάλισης ε, επιτρέπεται κάτι τέτοιο. Ε, πραγματικά εδώ αρνούμαστε θεμελιώδη δικαιώματα ε, και θα πρέπει να το επενθυμίσουμε αυτό. Κάτι ακόμα, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάνκα που έθεσε το ζήτημα του εθελοντικού ε, ταμείου συνταξιοδότησης ε, είναι ένα έτσι ε, λεπτό ζήτημα, το παρακολουθώ εδώ και καιρό. Το ταμείο αυτό το δημιούργησε το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο πήρε αυτή την απόφαση, έτσι. Και είπε στα μέλη, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ταμείο αυτό, εφόσον εσείς συνεισφέρετε μηνιαία πέρα από μια άλλη συνεισφορά του Κοινοβουλίου. Δύο τρίτα το Κοινοβούλιο και ένα τρίτο το κάθε μέλος του Κοινοβουλίου. Αυτό προέβλεπε ο κανονισμός και αυτό κάναμε. Όταν καθορίσαμε ποιο θα είναι το καθεστώς των μελών, εκεί αναφέρεται ρητά ότι αυτά τα όποια δικαιώματα έχουν προκύψει από αυτό το ταμείο θα παραμείνουν στο ακέραιο, χωρίς όριο. Δεν θέλω λοιπόν τώρα να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα ε, και να λέμε εδώ ότι κάποιοι προσπαθούν να αποτελεστούν μια κατάσταση ενώ είναι μια πρωτοβουλία του Προεδρείου ε, εδώ και χρόνια με τη στήριξη του συνόλου του Κοινοβουλίου. Έχουμε αναλάβει κάποιες δεσμεύσει. Όταν έχουμε αναλάβει δεσμεύσει πρέπει να τις σεβόμαστε. Αυτά, Πρόεδρε, ήθελα να πω και επιβεβαιώνω προ τον συνάδελφο τον κύριο Μάνκα ότι είμαστε στη διάθεσή του για να συζητήσουμε και να βρούμε τι καλύτερε δυνατέ λύσει ε, στα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκε. Μάλιστα, ευχαριστώ τον κύριο Ντεπρέ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ομαρτζή για την ΚΟΕ. Όμως, ε, όχι, δεν θέλει το λόγο ο κύριος Ομαρτζή. Ίσως ο κύριος Ταγόν θα μιλήσει για τους πράσινους. Ευχαριστώ. Ναι, να μιλήσω και για τους πράσινους αν θέλετε. Ε, για την ΚΟΕ, συγγνώμη. Ε, άμα θέλετε. Εδώ εκπροσωπώ όμως τη Χέλγα Τρούπελ που είναι η σκιώδης μας και μου ζήτησε να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ε, Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κύριο Μάνκα για τη σπουδαία του εργασία που βρίσκει ευρεία στήριξη. ανάμεσα στα επιπλέον και συμπληρωματικά στοιχεία μέσα στις τροπολογίες, πιθανό είναι να στηρίξουμε τα εξής, δηλαδή πλήρης ε, ε, μοιρασιά των ε, λειτουργιών. Αυτό είναι καλύτερα να το κάνουν οι επιτροπές, κάποια πράσινα στοιχεία για τις μεταφορές που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, αμφισβήτηση του ρόλου της DGCOM όσον αφορά την φύση της ε, ανακοίνωσης των προκαταρκτικών συμφωνιών, όπως ας πούμε για την οδηγία περί copyright και βεβαίως ε, θέματα διαφάνειας. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι συμφωνούμε με τον εισηγητή πως υπάρχει χώρος για εξοικονομήσεις και τροποποιήσεις όσον αφορά την πρόταση που είναι τώρα επιτάπητος. Τέλος, εγώ προσωπικά, τα δικά μου προσωπικά σχόλια είναι ότι θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Ντεπρέ για τα όσα είπε για την εκπροσώπηση του ομοσπονδιακού θεσμού σε διάφορες περιοχές και τους ε, επικόους. Είναι πρόβλημα Ίσως θα έπρεπε να είμαστε πιο σφιχτοί σε αυτή την γραμμή. Ωστόσο, ε, διαφωνώ με τον κύριο Τεπρέ για το Ταμείο Ιδιωτική Συνταξιδότηση. Είπατε ότι φτιάχτηκε από το Κοινοβούλιο και έχετε δίκιο. Η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου το υπερψήφισε αυτό. Από την άλλη πλευρά, όμω, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν ήταν τόσο έντιμη και καλή πρόταση αρχική επί της οποίας μετά ψήφισε το Κοινοβούλιο και περιλάμβανε τον κίνδυνο ενός ιδιωτικού κοινο, ε, ιδιωτικού ε, ταμείου. Δεν ήταν κοινοβουλευτικό και συνταξιδιωτικό ταμείο. Όταν λοιπόν το είδαμε πριν από ένα χρόνο ε, περίπου και κάτι παραπάνω για πρώτη φορά, Εγώ θα έλεγα ότι τα μέλη που συνέβαλαν σε αυτό το ταμείο θα πρέπει να αποζημιωθούν για το, δικό, για το κομμάτι αυτό. Τα υπόλοιπα όμως είναι ένας κίνδυνος που αναλαμβάνεις όταν έχεις να κάνεις με ιδιωτικά ταμεία του Λουξεμβούργου. Και τούτου λεχθέντος, όλοι κάποτε θα πάρουμε σύνταξη. Ίσως θα να τα πω άλλα, να τα πω αλλιώς. Σας ευχαριστώ. Τώρα μπορείτε όσοι θέλετε να πάρετε το λόγο. Η Έντερ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα θέλω να συγχαρώ τον κύριο Μάνκα για τις προτάσεις που μας υπέβαλε ε, είναι πολύ θετικές. Ε, έχουν, ε, έτσι κι αλλιώς ακολουθούν την γραμμή της ομάδας στην οποία ανήκουμε και οι δύο και συμφωνούμε με τα όσα έχουμε συζητήσει εντωμεταξύ σε αυτή τη θητεία και γι' αυτό θα βρούμε και συμφωνία με τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες. Συμφωνώ με τον κύριο Ντεπρέ που λέει ότι πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι στην έκθεση για το τι νούμερα θέλουμε να μειώσουμε στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου και μέχρι ποιο σημείου σημείο θέλουμε να προχωρήσουμε. Αυτό πρέπει να το έχουμε καθορίσει ανάμεσα στις ομάδες μέσω των διαπραγματεύσεων και εμείς, όπως είπα, θα, και θα στηρίξουμε την αύξηση του προϋπολογισμού γύρω από τον πληθωρισμό ή παρόμοιο ε, σε σχέση με το πόσο αυξήθηκε την προηγούμενο χρόνο, γιατί τα νούμερα έτσι δεν διαφέρουν πολύ. Δεν έχει γίνει τίποτα το έκτακτο που να, που να δικαιολογεί αύξηση περισσότερη από το κόστος της ζωής. Όσον αφορά τώρα μασάζε, αυτό είναι θέμα που έχει απασχολήσει στη διάρκεια αυτή τη στιγμή Είναι μια τεχνική δημοσιονομική όπου τα χρήματα που στο τέλος της χρήση δεν έχουν απορροφηθεί μπορούν να μετακινηθούν και να πληρώσουν άλλα πράγματα που έπρεπε να έχουν πληρωθεί. Αυτό είναι σωστό. Αυτό όμω που δεν μου φαίνεται σωστό είναι να ε, αν ας πούμε να μείνουν 100 ε, γραμμές χωρίς να απορροφηθούν ε, επίτηδες και να κρύβεται έτσι αυτό που, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ώστε να χρησιμοποιείται για τα ε, κτίρια. Ε, αυτό δεν μου φαίνεται σωστό. όχι το να χρησιμοποιούμε αυτά που πραγματικά μας περίσεψαν. Τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα έχουμε κάποια σημεία που, όπως αυτό που είπαμε για τις συντάξεις των APA. Δεν είναι φυσιολογικό όταν έχουν κάνει τη δουλειά τους για δύο θητείες, μόνο και μόνο για ένα διοικητικό λόγο και μόνο γιατί το 2014 γίνανε οι εκλογές ένα μήνα νωρίτερα και άρα δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τα δύο χρόνια ε, να μείνουν χωρίς αποδοχές. Ε, από ό,τι κατάλαβα έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω πως ο κύριος, ο κύριος Μάγκα σωστά το έθεσε για να μην τους ξεχάσουμε. Το ίδιο με τις αποζημιώσεις που, λάβουν οι βοηθοί, λαμβάνουν οι βοηθοί μας όταν πάνε σε αποστολές. Ζητήσαμε να είναι στο ίδιο επίπεδο όπως οι υπάλληλοι του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί ακριβώς οι δαπάνες είναι οι ίδιες, είτε είσαι ε, υπάλληλο είτε είσαι βοηθός. Το μόνο που πετύχαμε ήταν μια μικρή ε, ενημέρωση περίπτωση Δεν έχει γίνει όμως εξίσωση. Νομίζω πως αυτό πρέπει τώρα να γίνει, είναι η καλύτερη στιγμή, γιατί έτσι όταν θα ξεκινήσει η νέα θητεία, οι νέο εκλεγέντες βουλευτές θα γνωρίζουν ποια είναι τα κόστη και να μπορούν να προσαρμόσουν τις δαπάνες των γραφείων τους, έχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ε, στα χέρια τους. Για να μην αλλάζουν δηλαδή οι κανόνες του παιχνιδιού στη μέση της ε, θητείας. Και για να είναι όλοι στις ίδιες, τις ίδιες συνθήκες μόλις αρχίσει η νέα θητεία. Κάτι ε, ακόμα είναι τα απαραίτητα μέσα για να καταπολεμηθεί η παρενόχληση και τα θύματα του παρενόχλησης να μπορούν να βοηθηθούν να προβούν σε καταγγελία και όλα να διεκπαιρεωθούν έγκαιρα. Ο κύριος Μάνκα το ξέρει πολύ καλά ε, ότι δεν έχουμε το απαραίτητο και κατάλληλα ε, εκπαιδευμένο, καταρτισμένο προσωπικό για να κάνει αυτή τη δουλειά. Και τέλος, επεξηγήσεις ψήφου που ο κύριος Μάνκα προτείνει να το αλλάξουμε. Εγώ θα ήμουν πιο ριζοσπαστική. Θα έλεγα να καταργηθούν τελείως. Νομίζω πως έχει δίκιο όταν λέει ότι τελικά ε, έχουμε αρκετά μέσα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε γιατί ψηφίσαμε το τάδε ή το δίνα. Μπορούμε να το κάνουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων. Το Κοινοβούλιο θέτει στη διάθεσή μα ένα σωρό ε, υπηρεσίε οπτικοακουστικές και νομίζω πως ε, θα μπορούσαμε έτσι να κάνουμε μια σημαντική εξοικονόμηση εάν δεν είχαμε αυτή τη μια μισή ώρα επεξηγήσεων ψήφων καθημερινά με όλε τι υπηρεσίε διερμηνία σε όλε τι γλώσσε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή το κόστο δεν δεν δικαιολογεί τα ωφέλη που είναι προσωπικά ή ατομικά το να μπορεί κανείς δηλαδή να κάνει τις επεξήγησεις ψήφου. Αυτά λοιπόν δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστώ Έντερ και τώρα ο Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ προσυπογράφω τα όσα είπε ο συνάδελφος Γεράρ Ντεπρέ αλλά ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον συνάδελφο Μάνκα για τη δουλειά του. Καταρχάς, να το πω να αντισταθεί, να είναι δυνατός ε, απέναντι στο λαϊκισμό. Πολλές φορές ε, γίνονται ένα σωρό τέτοιες προσπάθειες ε, και ξέρουμε ότι ορισμένοι από αυτούς ε, προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη στη διάρκεια των προεκλογικών ε, περιόδων ε, για δαπάνες που είναι όχι μόνο νόμιμες αλλά και απόλυτα αιτιολογημένες. Εμείς ανέκαθεν στηρίζαμε αυστηρό προϋπολογισμό αλλά με τα επαρκή χρήματα. Ε, έχουμε διάφορες υπηρεσίες, έχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αν δεν τις έχουμε τότε η δημοκρατία θα χάσει αλλά και η ποιότητα της νομοθεσίας μας. Και αυτή η ε, νομοθετική αριστεία θα πρέπει να, ε, νομοθετική αριστεία θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ένας από τους στόχους μας. Να μην μιλάμε μόνο για το κόστος και ούτε είναι τόσο τεράστιο το κόστος. Το κόστος της κακής νομοθεσίας θα είναι πολύ μεγαλύτερο για τους πολίτες. Ε, γι' αυτό λοιπόν και συμφωνούμε κατά βάση με την πρόταση του εισηγητή. Είναι προφανές ότι όπου μπορούμε να αποταμιεύσουμε, να ξεκονομήσουμε βασικά, θα πρέπει να το κάνουμε. Γνωρίζοντας ωστόσο ότι για το Κοινοβούλιο, ας πούμε, για θέμα, όσον αφορά τα ποσοστά του τίτλου 5, Μειώνεται μάλιστα το ποσοστό σε σχέση με, τις άλλες, ε, με, τα, με τα, τους άλλους θεσμούς. Στον ευρωπαϊκό προπολογισμό το βάρος των θεσμών και της λειτουργίας τους αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 7% το ετήσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συχνά Έχουμε περάσει περισσότερο χρόνο, περνάμε μάλλον περισσότερο χρόνο μιλώντας για αυτό το 7% αντί να μιλάμε για το υπόλοιπο 93% που είναι ουσιώδες, για την αντιγωνιστικότητα της Ένωσης, για τη λειτουργία της Ένωσης, για τη βοήθεια ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για το Ταμείο Συνογής, ε, Εδαφικής Συνοχής και Οικονομικής Συνοχής. Άρα λοιπόν... Το, επό, το, το, παράδειγμα που πρέπει να δώσουμε σε όλα τα επίπεδα είναι, ε, το θέμα, είναι η διαφάνεια, απόλυτη διαφάνεια. Και μετά, σε σχέση με την ανάγκη που έχουμε πάντοτε να είμαστε άγρυπνοι, εμ, να είμαστε υποδειγματικοί και να προσπαθούμε να μειώνουμε όσο γίνεται περισσότερο τις απαραίτητες δαπάνες. Και αυτό κάνοντας ε, συνεργίες για να έχουμε εξοικονομήσεις. Προσπαθούμε πάντα με λιγότερα να τα πάμε καλύτερα. Λιτότητα, το μίνιμουμ που είναι απαραίτητο όμως γιατί είναι νομοθετική αριστεία θα πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Χωσέ Μανουέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Χάουαρντ. Δεν θα ήθελα να πω τίποτα αρχικά, αλλά ε, αναγκάζομαι από τα όσα ακούω. Για, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ήμουν στο Ηνωμένο Βασίλειο επικριτικός για το είδος των εγκαταστάσεων και τη χρηματοδότηση που δινόταν στα βουλευτές του Westminster για να κάνουν τη δουλειά τους αντιπροσωπεύοντας τους εκλογίστους. τους. Εγώ βρίσκω πως εδώ έχουμε κάποια από αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα βασικό επίπεδο χρηματοδότησης που επιτρέπει στους ευρωβουλευτές να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Και επίσης νομίζω ότι το να διατηρηθεί αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε πως τα διάφορα κρατημέλη έχουν διαφορετικές ε, ε, ε, συνήθειες, κουλτούρες και διαφορετικά μεγέθη περιφερειών. Δεν μπορούμε λοιπόν όλους να τους βάλουμε σε ένα καλούπι. Άρα λοιπόν η έννοια ότι πρέπει να περιορίσουμε τα μέσα που έχει ο κόσμος για να βάλουμε αυτή τη θέση ε, να τη δημοσιεύσουμε, να παρεμβαίνουμε εδώ ως απλά μέλη του Κοινοβουλίου, όχι ως πρόεδροι των Επιτροπών ή ως συντονιστές ή ως εκπρόσωποι, αλλά εν πάση περιπτώσει οι ευρωβουλευτές να βάζουν, να καταγράφουν τη θέση τους και να μπορούν έτσι να επικοινωνούν με το κοινό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην περιορίσουμε το ε, κοινοβούλιο στην ε, στους γλωσσολόγους ε, ή στους ειδικούς των γλωσσών. Πιστεύω πως είναι απαραίτητοι όλοι. Είναι απαραίτητοι για να μπορούμε να επικοινωνούμε μεταξύ τους. Το κόστος των γλωσσών είναι απαραίτητο. Ε, ο ο κόσμος στις χώρες μας πρέπει να μπορεί να καταλάβει τι γίνεται εδώ μέσα στη γλώσσα τους. Είναι ζωτική σημασία για τη δημοκρατική πρόσβαση και αν η Ένωση είναι σπουδαία, ε, νομίζω πως είναι το δικό μας δώρο προς τον κόσμο να δίνουμε ναι την γλώσσα μας τα αγγλικά ως lingua franca, αλλά δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική. Οι δικές μου προσπάθειες να επικοινωνήσω σε άλλες γλώσσες ας πούμε προσωπικά είναι ισχνές, αλλά εν πάση περιπτώσει ο κόσμος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται και ε, είναι μεγάλο πρόβλημα εάν προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις γλώσσες στο Ευρωκοινοβούλιο. Euh, euh, Ευχαριστώ. Αν θέλει κανεί άλλο το λόγο να σα πω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι εδώ τα άστρα είναι μαζί μα, μιας και το εισηγητή είναι και μέλος του Προεδρείου. Ε, θέλω να τον ευχαριστήσω λοιπόν. Φέτο ε, είχαμε την κοινοποίηση ε, του project αυτού και υποβολή του σχεδίου προπολογισμού στο Προεδρείο ταυτόχρονα. Ε, είναι μια καινοτομία. Θα πρέπει βεβαίως ε, να συμβαίνει αυτό κάθε χρόνο. Το γεγονό ότι είστε μέλος του Προεδρείου, κύριε Μάνκα, σας επιτρέπει να απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα, όπως το θέμα της ε, ε εκπροσωπικής μας, της διπλωματικής ανά τον κόσμο πρέπει να σα πω προσωπικά ότι η Ευρώπη δεν έχει αρμοδιότητες ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ήδη υπηρεσία εξωτερική δράση. Ε, εάν το Κοινοβούλιο θέλει και αυτό να έχει τι δικέ τη διπλωματικέ αντιπροσωπείε, όταν θα έρθουν οι συμπολίτε μα να, να μα ρωτήσουν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, πρέπει να μπορούμε να του απαντήσουμε. Να το αιτιολογήσουμε. Να αιτιολογήσουμε αυτέ τι δαπάνε διότι είναι δημόσιο χρήμα. Θα πρέπει λοιπόν να αιτιολογείται η διάθεσή του. Κύριε Μάνκα τώρα θα απαντήσετε στους συνδέλφους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που έκαναν. Τα κατέγραψα όλα και είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι τα πιο πολλά στοιχεία μπορούμε να τα επιλύσουμε από κοινού. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω όλος ιδιαίτερος, γιατί στο παρελθόν ασκήσατε μεγάλη πίεση, προκειμένου η έκθεση να περάσει από το Προεδρείο κατευθείαν στην Επιτροπή Προπολογισμού. Δεν χρειάστηκε να το φροντίσω αυτό, γιατί ο Γενικός Γραμματέας είχε ήδη προτιμάσει τη διαδικασία αυτή μεταξύ άλλων και χάρη στην πίεση που άσκησε ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα να απαντήσω στον συνάδελφο Χόρβατ. Το ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι βέβαια. Οι βουλευτέ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν στη γλώσσα του. Εγώ όμω θα ήθελα να τονίσω το εξή τις προφορικέ αιτιολογήσει ε, ψήφου, στι επεξηγήσει ψήφου. Εδώ νομίζω ότι μπορούν να γίνουν οικονομίε, δηλαδή να μιλάει ο κάθε βουλευτή στη γλώσσα του, αλλά να παρουσιάζεται αυτό στην εκάστοτε χώρα. Αλλά και δεν υπάρχει συζήτηση ουσιαστικά, διάλογο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει διερμηνία σε 24 γλώσσε. Αυτό κοστίζει υπερβολικά πολύ και ο κάθε βουλευτή μπορεί να έπαιξει την ψήφο του στη χώρα του, στη γλώσσα του, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να μεταφράζεται. Συμφωνώ με την άλλη. θα μπορούσαμε να τις καταργήσουμε και παντελώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να ακολουθήσουμε και μια βαθμία προσέγγιση. Σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να βάλουμε και να αναβάλουμε όλες τις ε, αιτιολογήσεις ψήφου στο τέλος, τέλος της Ολομέλειας, προκειμένου εκεί να επεξηγεί όποιο θέλει την ε, ψήφο του και στη συνέχεια βλέπουμε ποια ήταν τα επόμενα βήματα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Υπάρχουν γραπτά αιτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταχωρίζονται και πολλοί βουλευτές θέλουν να υποβάλουν ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παίρνουν ε, πόντους. Αλλά αυτές οι ερωτήσεις κοστίζουν πάρα πολύ. Και στην Επιτροπή το έθιξε το θέμα αυτό ήδη πριν από δύο χρόνια. Η Επιτροπή αυτή είχε συμφωνήσει μαζί μου προκειμένου οι ερωτήσει αυτέ προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην συγκαταλέγονται, να μην ε, συμπεριλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία. Γιατί αν δεν συμπεριλαμβάνονται στα στατιστικά στοιχεία, οι βουλευτέ θα έθεταν μόνο τι ερωτήσει τι οποίε πραγματικά ήθελαν να θέσουν και δεν θα έλπιζαν με τον τρόπο αυτό να πάρουν πόντου. Στην Επιτροπή Προπολογισμού συμφώνησαν μαζί μου οι συνάδελφοι. Στην Ολομέλη όμω δεν μπορέσαμε να το περάσουμε μία περαιτέρω μεταρρύθμιση, η οποία έγινε ωστόσο από το 2015 και μετά. Μειώσαμε κατά 9.000 ε, τις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι κάναμε εξοικονόμηση 6,3 δισεκατομμύρια. Αυτό ήταν μεγάλο πόσο, μεγάλη οικονομία, γιατί πολλές από αυτές τις ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι περιττές. Πολύ έθεξαν το θέμα του συνταξιδευτικού ταμείου. Συμφωνώ με τον κύριο Ντεπρέ. Χθε είχαμε συνομιλίες με τον κύριο Γκράχαμ Βότσον, ο οποίος ήδη έχει συνταξιοδοτηθεί και πλέον η ηλικία συνταξιοδότηση είναι 65 έτη και ο κύριος Γκράχαμ ε, Βότσον ουσιαστικά θα έμενε χωρίς καμία κάλυψη. Και αυτό το ενημερώθηκε δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη της συνταξιοδότησης. Δεν είναι δυνατόν να αλλάζουν αυτά τα πράγματα τόσο άμεσα. Αν αλλάζουν οι παροχές, οι συνταξιοδοτικές, αυτό θα πρέπει να το ανακοινώνεται δύο, πέντε χρόνια πριν την έναρξη της ισχύω ε, της αλλαγής αυτής. Ε, αυτός, για παράδειγμα, ο Ευρωβουλευτής θα χάσει μεγάλο πόσο από τη συνταξιοδότησή του. Δεν είναι δυνατόν να ενημερώνεται αυτό έτσι απλά δύο εβδομάδε πριν για το ραμασάζ. Αυτό. Από τότε που δουλεύω εδώ, προσπαθώ να ακολουθήσω την εξή προσέγγιση. Να γνωρίζουμε τι οικονομίε θα γίνουν το συντομότερο δυνατό. Αν για παράδειγμα πληρώνουμε νωρίτερα τα έξοδα για τα κτίρια, ουσιαστικά κάνουμε μεγάλη εξοικονόμηση των επιτοκίων. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν έγκυρος προγραμματισμός και έγκαιρη παροχή των πληρωμών. Αν ε, γλιτώνουμε λοιπόν τα επιτόκια, ουσιαστικά μπορούμε να γλιτώσουμε μεγάλα ποσά και τα ποσά αυτά που γλιτώνουμε από τους στόχους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάπου αλλού. Πολλοί ανέφεραν ότι θέλουν να έχουν στην διάθεσή τους συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φερνάντες. Χρειαζόμαστε αριθμητικά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελέγχω τακτικά. Και όταν γνωρίζω ότι κάθε χρόνο έχω ένα ποσό ε, που περισσεύει σε κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο, μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό ως ε, επιχείρημα για το μέλλον. Ότι εκεί μπορούν να γίνουν οικονομίες. Αλλά θα πρέπει να είμαι και σίγουρος ότι δεν θα προκαλέσω και προβλήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Στις 14 Μαρτίου, λοιπόν, θέλω να υποβληθούν συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Έχω ήδη συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία στα εγγραφά μου, αλλά θα ήθελα να είμαι σίγουρος ότι τα στοιχεία αυτά είναι ρεαλιστικά. Έχω όμως όκτα ψήφια αριθμητικά στοιχεία εδώ σε ό,τι αφορά τις οικονομίες που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό δεν το λέω με διαθέσει, αλλά θα σας τα επιβάλλω αυτά, θα σα τα επιβάλλω σε μετέπειτα χρονική στιγμή, όπως σας είπα. Αναφέρθηκε και το θέμα της ομοσπονδιοποίησης. Ε. Οι αντιπροσωπείες δεν ε, ιδρύονται σε όλα τα κομμάτια του κόσμου, σε όλα τα τμήματα του κόσμου. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και στις, ε, στη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων αργότερα το Μάρτιο. Να σας ευχαριστήσω όλους σας για την ανταλλαγή απόψεων και προσβλέπω στις μελλοντικέ ε, συναντήσεις με τους κοιόδες εισηγητές σας ε, εύχομαι και μας εύχομαι ένα καλό προϋπολογισμό, ο οποίος να αντέχει στους κλειδονισμούς, αλλά και παράλληλα να χρηματοδοτήσει όλα όσα χρειάζεται να χρηματοδοτηθούν. Να μην αναστέλλονται δηλαδή έργα χωρίς να υπάρχει λόγος ουσιαστικός. Merci, monsieur le rapporteur. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Το σχέδιο προπολογισμού του Κοινοβουλίου, λοιπόν, ελπίζουμε να είναι το καλύτερο δυνατό. Σα έχουμε εμπιστοσύνη. Βεβαίω θα πρέπει να είμαστε αυστηροί και λυτοί. Είμαστε η Επιτροπή Προπολογισμού και πρέπει να προτείνουμε δαπάνες, μείωση δαπανών για να μην μας μπορεί να μας κανείς για κακή χρήση των δημοσίων δαπανών δεν φορολογούμε εμείς βέβαια, όμως τους φόρους τους ψηφίζουν οι συνάδελφοί μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια και σύμφωνα με τη συνθήκη διατίθεται τα χρήματα αυτά, μέρος των χρημάτων στους ευρωπαϊκούς προπολογισμούς, οπότε λογοδοτούμε για το πόσο αυστηροί είμαστε σε ό,τι αφορά τη χρήση των δημοσίων πόρων. Λοιπόν, κλείνουμε με το σημείο αυτό. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Το χρονοδιάγραμμα είναι το εξής. 13 Μαρτίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 13 Μαρτίου στη μια το μεσημέρι. 18 Μαρτίου θα έχουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για να εξετάσουμε τις ε, τροπολογίες. 25 Μαρτίου θα έχουμε την έγκριση του σχεδίου του κυρίου Μάνκα που θα περιλαμβάνει και τις ε, τροπολογίες και 27-28 Μαρτίου στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε το σχέδιο έκθεσης. Μου λένε ότι επειδή οι προθεσμίες αυτές είναι πολύ σφιχτές, ε, θα είναι στα αγγλικά οι τροπολογίες. Κάτι βεβαίω που δεν συνάδει με αυτό που πολύ σωστά είπε ο κ. Χάουαρτ προηγουμένως. Και τώρα θα ακούσουμε τους, αυτούς που εκπώνησαν μια μελέτη που ζητήθηκε από την θεματική ε, ομάδα των, της ομάδας προπολογισμού για να δούμε κατά πόσο η αρχή της όρτας των δύο φύλων γίνεται σεβαστή στα πλαίσια της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης. Αυτή, τη, αυτή η μελέτη Πρόκειται για επικαιροποίηση της μελέτης του 2015. Την εκπώνησε μια ομάδα ε, των κυρίων Μπλομέιρ και Σάνθ ε, υπό τη διεύθυνση του κυρίου Φιράτ Τσεντίζ. Ε, πρόκειται για μια μελέτη που εγγράφεται στο ευρύτερο σχέδιο δράση για την ισότητα των δύο φύλων που έκανε την Επιτροπή Προπολογισμού. Η κυρία Γκάρτια Θάβαλ και η κυρία Σούλιν είναι οι δύο εισηγήτριες για την Επιτροπή μας. Δώσα το λόγο πρώτα στον Δόκτωρ Τσεντίζ που θα μας παρουσιάσει εν συντομία τα συμπέρασματα της έκθεσης αυτή. Τον λέω εν συντομία 10 λεπτά εννοώ, έτσι. Um, thank you very much. It's a... Ευχαριστώ, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ. Το όνομα μου είναι Φυρά Τσεντίζ ε, και εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ ε, και το 2015 είχα έρθει εδώ δύο φορές να παρουσιάσω την προηγούμενη έρευνα. Ελπίζω να δούμε τώρα και κάποια πρόοδο, που, την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε ό,τι αφορά το θέμα της όντας των δύο φύλων στην Ένωση. Λοιπόν, ε, υπάρχει η άποψη Κάποιοι θεωρούν ότι σημαίνει ότι πρέπει να διαθέτουμε χρήματα για τι ισότητε των δύο φύλων ε, στον προπολογισμό. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Οι άντρε και οι γυναίκε ε, ε, γενικότερα επηρεάζονται διαφορετικά από τι διάφορε δημόσιε δαπάνε, ανάλογα με το που βρίσκονται κοινωνικά, είναι διαφορετικέ οι απαιτήσει και οι προπολογισμοί που αλλά το λαμβάνει υπόψη αυτό δεν ε, συνεισφέρουν μόνο στην ισότητα των δύο φύλων, αλλά και σε άλλες αξίες, λογοδοσία, δημοκρατία, Γι' αυτό λοιπόν οι διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων και τα Ηνωμένα Έθνη, έχουν ζητήσει να υπάρχει αυτό το gender budgeting εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει η πλατφόρμα για τη δράση του Πεκίνου των Ηνωμένων Εθνών που ζήτησε από όλα τα μέλη της να ακολουθήσει μία προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τα δύο φύλλα στην, εκπόνηση του προπολογισμού. Υπάρχει μια συνολική ε, επίση υποχρέωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τι των δύο και αυτό περιλαμβάνει και τον προπολογισμό. Οπότε δεν χρονίζω να χρειάζεται να αλλάξει κάτι νομοθετικά για να εισαγάγουμε αυτήν την, ε, αυτό το καθήκον, αν θέλετε, ε, για να λαμβάνετε υπόψη το ζήτημα στον προπολογισμό. Το 2015 στη μελέτη μας είχαμε εξετάσει το θέμα της όντως των δύο φύλων ε, στους του 2014 και του 2015 καθώς και στα πλαίσια του προηγούμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και οι, ε, οι δεσμεύσει υψηλού επίπεδου για την ισότητα των δύο φύλων δεν ακολουθήθηκαν με συνέπεια και συστηματικά στην εφαρμογή στη συνέχεια. Στήσαμε λοιπόν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Κομισιόν από κοινού να αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό με κάποια κοινή δράση. Στην παρούσα μελέτη μελετήσαμε τις ενδεχόμενες βελτιώσεις από το 2015 έως σήμερα υπό το φως των ετήσιων προπολογισμών αλλά και του επόμενου πολιτός δημοσιονομικού πλαισίου. Και αυτό το κάναμε με βάση έρευνες και συνεντεύξεις με έξι γενικές διευθύνσεις που είναι υπεύθυνε για τους τομείς πολιτικής που καλύπτουμε. Όπως ξέρετε υπάρχει μια ψήφιση το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν χρειάζεται να το επαναλάβω η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και το ζήτημα αυτό έχει, δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού προγράμματο. Είναι πραγματικά, είναι πραγματικά λυπηρό αυτό, διότι είμαστε ακόμα μακριά από το να πετύχουμε την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Και σε ό,τι αφορά του νέου κανονισμού που εγκρίθηκαν ε, για να μεταρρυθμιστεί το πρόγραμμα δαπανών, ε, ούτε εκεί βλέπουν να υπάρχει μια συνεπής προσέγγιση που να σέβεται και να δέχεται την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων ως οριζόντια αρχή. Το έχουμε πει και στο παρελθόν και στην προηγούμενη έκθεση. Δηλαδή, ε, κάτι που μας λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι το πρόγραμμα DAFNE που είναι ένα πολύ επιτυχές πρόγραμμα για να αντιμετωπιστεί η βία η ενδοκογενειακή. Ε, ουσιαστικά είναι στο τρίτο επίπεδο και πρέπει να ανταγωνιστεί πολλές και πολλά και πολλά άλλα προγράμματα. Πολύ μικρή πρόοδος λοιπόν από τότε που έγινε η μελέτη μας το 2015. Πολύ λίγα πράγματα. Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων εξακολουθεί να μην είναι θεμελιώδης αρχή που να αναγνωρίζεται με συνέπεια στον προπολογισμό τη Ένωση. Αυτό που διαπιστώσαμε στι συνεντεύξει είναι ότι οι γενικέ διευθύνσει τη Κομισιόν δεν έχουν μια συνεπή κατανόηση του τι σημαίνει ο προπολογισμό που λαμβάνει υπόψη τα δύο φύλλα. Ε, δεν καταλαβαίνουν πώ αυτό θα γίνει στην καθημερινή εργασία των ευρωπαϊκών οργάνων. Βεβαίω έχουμε αντιμετωπίσει κάποια θετικά στοιχεία όπω το ΆΙΓΕ, η ΆΙΓΕ που έκανε τρει μελέτε ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε μια βάση πραγματογνωμοσύνη και μια βάση μεθοδολογία για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει έναν προπολογισμό που να λαμβάνει υπόψη τα δύο φύλλα. Υπάρχουν πλέον αρκετέ πληροφορίε, αρκετέ εμπειρίε που να υποστηρίζουν την, την να δράση στον τομέα αυτών εφόσον χρειαστεί. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του 2017 για το ζήτημα αυτό, καθώ και η Επιτροπή Προπολογισμού του 2018 στο σχέδιο δράση για την ισότητα των δύο φύλων, μα δίνουν και αυτά ελπίδα, μας δίνουν και αυτή η ελπίδα, διότι δεν είναι μόνο η Επιτροπή Γυναικών που ασχολείται με αυτό, ε, υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ διαφόρων επιτροπών και υπάρχει μια βούληση γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δοθεί έμφαση στο θέμα αυτό. Ε, με βάση όλα αυτά, οι συστάσεις μας, οι συστάσεις κλειδιά που είναι με αυτές του 2015 είναι οι εξή. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής για την ισότητα των διαφύλων πρέπει να γνωρίζεται ε, σε μακροοικονομικό επίπεδο όταν μιλάμε για μακροοικονομικό επίπεδο, εννοούμε τι γενικέ οικονομικέ πολιτικέ, ε, η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και βεβαίω υπάρχει και πολιτές, το, πολιτισμο το δημοσιονομικό πλαίσιο, καθώ και ο ετήσιο προπολογισμό, δηλαδή μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Το συστήνουμε αυτό διότι αν η ισότητα των δύο φύλων ε, έχει παραβλεφθεί, παραδείγματο χάρη στι μακροοικονομικέ πολιτικέ, είναι πολύ δύσκολο μετά τον ετήσιο προπολογισμό να το διορθώσουμε. Κάτι το οποίο δηλαδή έχει αγνοηθεί μακροπρόθεσμα. Η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων πρέπει να είναι πολιτικό στόχο σε όλου του τίτλου του προπολογισμού τη Ένωση, να υπάρχει μια συνεπή προσέγγιση και όλε οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό πρέπει να υπόκεινται σε gender mainstreaming. Αυτό είναι ένα καθήκον το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό σε όλε τι δράσει που λαμβάνουν χρηματοδότηση από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πρέπει να υπάρχουν δείκτε που να σχετίζονται με τα δύο φύλλα και να εγκρίνονται, να εφαρμόζονται στα πλαίσια της επιλογής των project αλλά και στην αξιολόγησή τους. Θα πρέπει να ακολουθούνται αυτές οι αρχές κατά τον, την, το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του προπολογισμού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κοινή δράση από την Κομισιόν, το Συμβούλιο και την Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μεταξύ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλε τι πλατφόρμε στη διάθεσή του και την Ολομέλεια, έτσι ώστε συνεχώ να, να μιλάει και να ζητάει περισσότερη ενισότητα μεταξύ των δύο φύλων και στου προπολογισμού ιδιαίτερα στις συζητήσεις στην Ολομέλεια, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ε, στην συζήτηση για την απαλλαγή, στη συζήτηση για τον προπολογισμό, γιατί εκεί είναι εκεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί τα μέλη του Κοινοβουλίου έχουν δυνατότητα να θέσουν ερωτήματα, να θέσουν το ζήτημα αυτό και να λογοδοτήσει η Κομισιόν. Θέλω να ζητήσω λοιπόν από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δημιουργήσουν μια συμμαχία για το ζήτημα αυτό και να δώσουν έμφαση ε, ιδιαίτερα στην Ολομέλεια. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο έγγραφο ο προπολογισμό, είναι πολλά αυτά που πρέπει να συζητηθούν, δεν υπάρχει αρκετό χρόνο. Οι διαδικαστικοί κανόνε ορισμένε φορέ ε, περιορίζουν τι συζητήσει, αλλά είναι πολύ σημαντικό και στην Ολομέλεια τα θέματα αυτά να τεθούν και να συζητηθούν. Κάπου εδώ τελειώνει η παρουσία μου, η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ε, κοινωνία και την εισήγηση. Το λόγο τώρα θα πάρει η Εντέρ Καρδία Ζαπάλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για όλες αυτές τις πληροφορίες και για την μελέτη που ε, μας δώσατε. Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε ε, γιατί, λίγο για την ε, παρουσίαση αυτής της έκθεσης. για να είμαστε κοντά στις 8 Μαρτίου είναι ένας, μια μέρα, μια επέτειος, μια μέρα που κατεβαίνουμε στους δρόμους και μάλιστα αυτό που είναι θετικό είναι ότι οι περισσότεροι άνδρες κατέβηκαν στους δρόμους ενώ παλιότερα περνούσε εγκόγνητο η μέρα αυτή και ελπίζουμε πως και αύριο θα γίνει αυτό. Και βεβαίως όταν βλέπουμε τα αποτελέσματα της ε, μελέτης ε, που ακριβώς αυτά είναι τα λόγια που είπε ε, η, η συγγήτρια, βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρή η πρόοδος, αν έγινε καν πρόοδος. Πραγματικά θα πρέπει να δούμε ε, ότι δεν έχουμε προχωρήσει σε αυτό το θέμα σχεδόν και ε, στην πολιτική ε, και στο mainstream είναι με το θέμα και του περιβάλλοντος. Το ίδιο συμβαίνει. Δεν είναι δύο θέματα άσχετα μεταξύ τους, αλλά δυστυχώς είδαμε ότι υπάρχουν δεσμεύσεις και από την άποψη ε, του προπολογισμού γίνανε διεθνείς συμφωνίες όπως η διάσκεψη του, του Παρισιού και την πολιτική ισότητα των φύλων. Όμως και ένταξη αυτής μέσα στον προπολογισμό βλέπω να μην γίνονται αρκετά. Δεν προχωράμε λοιπόν αρκετά, αλλά φτάνουμε και έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Και γι' αυτό ήταν ενδιαφέρον ε, το τι λέει αυτή η μελέτη. Έχουν καταγραφεί όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και πολύ συχνά η αδυναμία που έχουμε στους θεσμούς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να προωθήσουμε τα θέματα αυτά. Είναι αλήθεια και είναι αλήθεια για την ε, παρουσίαση αυτής της έκθεσης. Το Ινστιτούτο της Γυναίκας έχει κάνει διάφορες μελέτες και έχει δείξει πως είναι δυνατόν είναι δυνατόν, ε, δεν είναι τόσο περίπλοκο, ε, υπάρχουν πληροφορίες επαρκής και είναι δυνατόν να γίνει, είναι εφικτό. Ε, και αυτό με έκανε να προβληματιστώ, γιατί όταν χρειάστηκε να υπερασπιστώ πολιτικές για τα φύλλα και βέβαια προπολογισμού, πολύ συχνά μου έλεγαν «Α, δεν ξέρουμε, αχ, είναι δύσκολο, αχ, έχουμε άλλες προτεραιότητες». Κάθε φορά φαίνεται ότι η πολιτική της ισότητας και οι προπολογισμοί με εστιασμό στο φύλλο είναι στην ουσία η, η άκρη, η τελευταία στροχός της αμάξης. Δηλαδή κάνουμε πρώτα όλα τα άλλα και στο τέλος αν βρούμε χρόνο και χρήμα, <clears throat> εντάξει. Όμω ε, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερε προτάσει και συστάσει από πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου για το πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπορέσουμε να ε, πάμε καλύτερα στην επόμενη θητεία, να δώσουμε μια νόθηση και ε, την πολιτική του φίλου πραγματικά να την καταστήσουμε οριζόντια, να διαπερνά όλες τις άλλες πολιτικές. Έχουμε λοιπόν εδώ κάτι προτείνει και στο ε, δημοσιονομικό πλαίσιο η, αρχικά δεν ήταν προτεραιότητα, εμείς όμως το μετατρέψαμε σε προτεραιότητα. Ποια πιο συγκεκριμένα μέσα όμως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και εδώ νομίζω πως έχουμε πρόβλημα ενημέρωση, ε, μάλλον κατάρτισης εμείς, οι βουλευτές. Γιατί δεν ξέρουμε πολύ καλά τι, τι πρέπει ακριβώς να κάνουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να κατέβουμε ε, ε, στο, ε, στο πεδίο που πρέπει και να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πιστεύω λοιπόν πως πρέπει ως Κοινοβούλιο να κάνουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει ή που δεν έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω πως κάτι τέτοιο λοιπόν θα ήταν πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τομά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω. Είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Ε, καθώς μάλιστα το Κοινοβούλιο, όπως το ξέρετε, ψήφισε διάφορες ε, θέσεις για το μελλοντικό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, ε, για τις οποίες ζητάμε να γίνει επαλήθευση του προϋπολογισμού για την ισορροπία ανάμεσα στην ε, χρήση των ε, εργαλείων που έχουμε και όπως είπε και η κυρία Καρδιαζαμπάλ μόλις ε, χρειαζόμαστε ελεκτικά εργαλεία αλλά και εφαρμοστικά εργαλεία και ίσως εκεί ε, θα πρέπει να εστιαστεί το αίτημά μας αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν σε όλα όσα ψηφίσαμε, και αυτό το λέω για να δώσω ίσως κάποιες κατευθύνσεις, όταν ψηφίσαμε λοιπόν για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο λέει σαφώς ότι αυτή η αναθεώρηση ενδιάμεση θα πρέπει να ε, παληθεύσει την εξέλιξη του gender budgeting και ότι σε σχέση με το αποτέλεσμα αυτής της επαλήθευσης ε, τότε μπορούμε να τροποποιήσουμε και, αυτή και αυτό είναι και το νόημα της υποχρεωτικής αναθεώρησης, ότι μπορούμε και οφείλουμε να τροποποιήσουμε τα μελλοντικά προγράμματα, ή εν πάση περιπτώσει την κατανομή των μελλοντικών προγραμμάτων. Είναι αλήθεια ότι για την ώρα είναι γραμμένο κάπως πιο θεωρητικά, Αυτή η υποχρεωτική αναθεώρηση ενδιάμεση θα ήταν η κατάλληλότερη στιγμή για ε, μια ενδεχόμενη αλλαγή πορείας, αλλά θα πρέπει πολύ σωστά να προετοιμάσουμε τα ε, εργαλεία που θα έχουμε στη θέση μας. Και εδώ, όπως είπε η Έδερ, δεν το έχουμε αυτά. Α, λοιπόν, δεν είναι το Κοινοβούλιο που θα πρέπει να ορίσει ε, τα εργαλεία, είναι η Κομισιόν, αυτό λέει και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή να προετοιμάσει τα εργαλεία για αυτή την αξιολόγηση, αλλά επίσης και για αυτήν την αλλαγή πορείας και προσανατολισμού υπό τη μορφή των προγραμμάτων της Κομισιόν. Δεν είναι μόνο η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου βέβαια που θα ρυθμίσει το σύνολο των προβλημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό να έχουμε αυτή την πρώτη αξιολόγηση. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί λοιπόν και να μην ε, κάνουμε μόνο δηλώσεις, είναι απαραίτητο να έχουμε εφαρμοστικά μέσα και επαλήθευσης, μέσα επαλήθευσης και γρήγορη αξιολόγηση γιατί δεν μπορούμε κάθε φορά να κάνουμε μια αξιολόγηση στατικική, λεπτομερή κτλ. Χρειαζόμαστε μέσα, μέτρα, ε, μάλλον εργαλεία γρήγορης αξιολόγησης και μέσα προσανατολισμού στην εφαρμογή των πολιτικών. Σας ευχαριστώ. Ε, αυτό είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου θα αποτελέσει κεντρική ε, σημασία, οπότε καλύτερο είναι να επιταχύνουμε για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των πολιτών. Ε, δεν ζητάει κάποιος άλλος το λόγο. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να, σας, να μοιραστώ μαζί μου τις απορίες μου. Ε, βεβαίως εκτιμώ ιδιαίτερα την Αντέρα και ενθάρρυνα την πρωτοβουλία Πώς μπορεί κανείς να βάλει στον προπολογισμό την ισότητα των φίλων όμως. Περιμένω πολλά από τις διαδοχικές ε, εκθέσεις και από τη στιγμή που είπαμε ότι επί της ουσίας δεν μεταφράζεται στον προπολογισμό, θα ήθελα να μου πείτε δύο-τρία συστάσεις συγκεκριμένες. Δηλαδή, αν εσείς έπρεπε να κάνετε το προπολογισμό, τι θα κάνατε ώστε να σεβαστείτε την ισορροπία των φύλων. Γιατί κάθε χρόνο ψηφίζουμε προϋπολογισμό. Και όλοι μας ε, μεριμνούμε και προσέχουμε την ισότητα των φυλών. Όμως συγκεκριμένα όταν λέτε ότι δεν υπάρχουν αρκετά μέτρα ώστε να μεταφράσουν την αρχή αυτή σε, στον προπολογισμό, πείτε μας δύο-τρεις συγκεκριμένες προτάσεις, αν θέλετε, που θα πρέπει να μπουν στον προπολογισμό μας. Έχετε το λόγο. Okay, thank you very much for the... Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις, γιατί όλες ε, ουσιαστικά προς την ίδια κατεύθυνση στρέφονται. Θέλετε να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο και να σας μιλήσω για εργαλεία. Και το τι θα μπορούσαν να κάνουν το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα. Προκειμένου να καταστεί αυτό μια πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την ε, θέτετε. Να σας πω το εξής καταρχάς. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ περίπλοκο αυτό, ιδέα, αυτή η διάσταση του φίλου στον προπολογισμό. Ουσιαστικά δεν είναι πάρα πολύ περίπλοκο όμω. Αυτό που σημαίνει είναι ότι όλοι μα, άντρε και γυναίκε, εξελίσσουμε την κοινωνία μας και αντιμετωπίζουμε με διαφορετικό τρόπο την κοινωνία. Αυτό το βλέπετε και στις ε, προσωπικές σας εμπειρίες, φαντάζομαι. Αντιμετωπίζουμε διάφορους περιορισμούς, εμπόδια, ανάλογα με την προσωπική μας εξέλιξη ως άτομα σε ό,τι αφορά τις ικανότητές μας, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευσή μας, την πρόσβαση στον εργασιακό κλάδο, στις πολιτικές πλατφόρμες, σε λοιπές πλατφόρμες, σε ό,τι αφορά τη λήψη αποφάσεων και όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πολλά και διάφορα. Αναπτύσσουμε λοιπόν αυτή την ευαισθησία και την εντάσσουμε και στις καθημερινές μας εργασίες. Ε, αυτό μπορεί να μην το κάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτε, αλλά εγώ το κάνω πάντα σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Πάντα εξετάζω αυτή τη διάσταση. Και ξέρω ότι πολλοί από εσά κάνουν το ίδιο στι συζητήσει αυτέ. Το 2019 και σε προηγούμενε συζητήσει εστιαστήκαμε ιδιαίτερα στο θέμα τη ασφάλεια και τη μετανάστευση, καθώ και τη οικονομική και νομισματική ένωση. Περίμενα λοιπόν κάποιον να θέσει και το θέμα του φύλου, τη διάσταση του φύλου σε ό,τι αφορά τα στοιχεία αυτά γιατί αυτά τα θέματα έχουν να κάνουν πάρα πολύ με το φύλλο. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που κατατεκνύουν ότι οι οικονομικές πολιτικές και η λιτότητα πλήττουν τις γυναίκες πολύ πιο βαριά από ότι τους άντρες. Όχι μόνο επιτυχάνουν τις δουλειές, τις δουλειές τους σε θέσεις παροχής υπηρεσιών, αλλά γιατί και το κράτος ουσιαστικά αποσύρει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη φύλαξη των παιδιών και τελικά οι γυναίκε είναι αυτέ που μένουν πίσω να φροντίζουν τα παιδιά, του αρρώστου, στο σπίτι. Και έτσι υπάρχει μια μετατόπιση δυνάμεων. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία να τα λάβουμε υπόψη σε καθημερινέ δραστηριότητε, ω άτομα, ω θεσμικά όργανα. Αν θέλετε να δούμε τα πράγματα πιο λεπτομερώς, έχουμε αναπτύξει ένα μια καλή εργαλειοθήκη για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα τέτοια. Στις καθημερινές δράσεις μας. Είναι πολύ γενική αυτή η, πρόταση, η οποία όμως μπορεί να δημορφωθεί με τεχνικούς όρους και να ενταχθεί στα πλαίσια του προϋπολογισμού. Όποιο είναι υπεύθυνο για τον προπολογισμό θα πρέπει να καταρτήσει σχετικού δείκτε για τα φύλλα. Τα κράτη-μέλη το κάνουν αυτό, αλλά επιδεικνύουν αφέλεια. Για παράδειγμα, στην Αυστρία είναι θέμα συνταγματικά κατοχυρωμένο το θέμα της ισότητας των φύλων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να διδαχθούμε από τέτοια παραδείγματα ή σε κάποιες χώρες Όταν παρουσιάζεται ένα νέο νομοσχέδιο, θα πρέπει να παρουσιάζεται και η διάσταση του φύλου και η επίδραση στα φύλλα. Από αυτό λοιπόν μπορούμε να διδαχτούμε. Αλλά για παράδειγμα μπορούμε να ζητήσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτήσει τέτοιους δείκτες για το πώς οι πολιτικές που προτείνει επηρεάζουν τη διάσταση του φύλου στην εκπαίδευση, στη μετανάστευση και παντού. Και επίσης στην έκταση περιλαμβάνονται κάποιες συγκεκριμένε προτάσεις σε ό,τι αφορά διάφορα προγράμματα που χάσανε ε, την ε, χρηματοδότησή τους και τώρα ανταγωνίζονται άλλα προγράμματα και τίθεται το θέμα όχι μόνο της ε, ισότητας του φύλου, αλλά και γενικά της διαφάνειας της νομοσχεδίας. Θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι οι γυναίκες πάντα οι χαμένες. Πολλά λοιπόν μπορούν να γίνουν σε τεχνικό επίπεδο και μη, αλλά το βασικό πόρισμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ευαισθητοποίηση σε ό,τι αφορά τη διάσταση του φίλου, σε ό,τι αφορά τις καθημερινές μας δραστηριότητε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Ζόλτεξ θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η 8η Μαρτίου είναι η μέρα διαμαρτυρίας που θα βγει ο κόσμος στους δρόμους. Δεν ξέρω τι γίνεται στις χώρες σας, αλλά στην Πολωνία ήθεστε την ημέρα εκείνη να επιδεικνύουμε την ε, αγάπη και το σεβασμό μας προς τις γυναίκες. Ενδεχομένω για άλλε χώρε αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να βγει ο κόσμο στον δρόμο να διαδηλώσει. Δεν είμαστε. Δεν είμαι πολύ καλό ε, στα φεμινιστικά. Αλλά αυτό που πιστεύω είναι ότι όλες οι γυναίκες θα... Όταν, μάλλον, οι γυναίκες προσπαθούν να είναι άντρες και οι άντρες προσπαθούν να εκτελέσουν τις, ε, ε, τα καθήκοντα των γενικών, ε, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Θα προτιμούσαν να είναι οι γυναίκες γυναίκες και οι άντρες άντρες. Οι γυναίκες είναι χαρούμενες όπως είναι και σας παρακαλώ λοιπόν να μην εξαναγκάζουμε τον κόσμο να αλλάξει ρόλο. Να μην ε, προσπαθήσουμε δηλαδή να εξαναγκάσουμε και τις γυναίκες που είναι ευχαριστημένες στο ρόλο τους ως γυναίκες να αλλάξουν και να είναι ε, άντρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ζόλτεκ εξέφρασε την προσωπική του άποψη στο πλαίσιο της Πολωνίας. Ε, Η κυρία Presidente, ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Από πού να αρχίσω. Εμπάσχευτος, ο κύριο Ζόλτεκ ε, δεν πρέπει να έχει και μεγάλες σχέσεις με ενώσεις γυναικών. Μια γυναίκα δεν θέλει να πάρει τη θέση του άντρα και ο άντρας τη θέση μιας γυναίκας. Δεν υπάρχουν καταρχήν δουλειές για άντρες και δουλειές για γυναίκες. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε. Εδώ υπερασπιζόμαστε την ισότητα των των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ο καθένας να μπορεί να είναι ελεύθερος να επιλέξει τι θέλει να κάνει, σε τι θέλει να αφιερωθεί και τι χρόνο θέλει να αφιερώσει στη δουλειά του, στην οικογένειά του και οπουδήποτε αλλού. Αυτή, αυτό είναι ένα από τα αιτήματα. Και όντω στη χώρα μου, στις 8 Μαρτίου, ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο. Και ευτυχώ κάθε φορά όλο και περισσότερε γυναίκες και άντρε βγαίνουν στον δρόμο. Πέρυσι, μάλιστα, ε, είχαμε μια από τι μεγαλύτερε διαδηλώσει στην Ισπανία. Σε τόσε πόλει και χωριά ε, δεν έχει γίνει αυτό εδώ και πολύ καιρό και για κάτι θετικό μάλιστα και όχι όπως τις 11 Μαρτίου του 2004 με τις τρομοκρατικέ επιθέσει. Για κάτι θετικό λοιπόν, για ένα θετικό λόγο κινητοποιηθήκαμε σε πόλεις και χωριά. Όπως και να έχουν τα πράγματα, συστήνω στον κύριο Ζόλτεκ να έρθει σε επαφή με τις ενώσεις γυναικών για να καταλάβει κάπως καλύτερα ποιες είναι, ε, ποια είναι τα αιτήματα. Διότι δεν πρόκειται για κάποια μάχη μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι μια κοινή μάχη, ένας κοινό αγώνας για να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκρέσλε, έχει το λόγο. Είμαι και πρόεδρο τη Ένωση Γυναικών στην περιοχή μου και εκπροσωπώ 14.000 γυναίκε στην περιφερειά μου και θα ήθελα να το επιστήσω αυτό το θέμα στον κύριο ε, Σόλτε. Αν δεν μπορεί να καταλάβει τα ε, γυναικεία θέματα, α καταλάβει τα ανδρικά θέματα. Οι άντρε ε, ζουν πιο ε, λίγο από ότι οι γυναίκε, με πιο ανθυγινό τρόπο, αντιμετωπίζουν πιο πολλά προβλήματα. αυτή η τάση να καταστρέψουν τη ζωή τους ε, χωρίς να αυτοκτονούν, θα πρέπει να μας κάνει να ρωτηθούμε από πού προέρχονται αυτές οι τάσεις. Γιατί σε τελική ανάλυση ε, δεν θέλουμε να έχουμε τις γυναίκες μόνους τους ε, να πολεμούν, να το διευκρινίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τωμά. Εν συντομία παρακαλώ. pense que je... Monsieur Viotti. Oui, non, là, Ναι, τα όλα κάτω. Εγώ σε θα είμαι πολύ σύντομη, Πρόεδρε. Να πω απλώς, όπως είπαν και δύο συνάδελφοι, το θέμα είναι η ισότητα. Δεν θέλουμε να πάρουμε από το ένα να δώσουμε στον άλλον. Εγώ είμαι πολύ φεμινίστρια. Α, έφυγε. Ε, δεν ξέρω, όχι δεν έφυγε. Ε, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε ότι έχω γίνει άντρα, αλλά αύριο θα είμαι στη Βαρσοβία και θα διαδηλώσω με τι φεμινιστικέ οργανώσει τι πολωνικέ. Φαντάζομαι ότι δεν θα είστε εκεί. Κρίμα, διότι το θέμα τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν είναι ένα θέμα που αφορά τι γυναίκε. Αφορά το σύνολο τη ανθρωπότητα. Σα ευχαριστώ. Donc, euh, nous avons une communication. Μάλιστα έχουμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση. Ξέρουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Ε, θα μας βοηθήσετε όμω, κυρία μου ε, να μας δώσετε συστάσεις πιο συγκεκριμένε. Γιατί ομολογώ ότι κάτι μου λείπει. Τι σημαίνει ένας προϋπολογισμός ο οποίος ανταποκρίνεται στην απέτηση αυτή ισότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών δεν έχω την εντύπωση στις εργασίες μας ε, το παραμελούμε αυτό. Προφανώς υπάρχει υπερθόριο βελτίωσης. Ε, θα, σύντομα στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε για σημαντικές, ε, σημαντικά αξιώματα. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ένα μέλος της Επιτροπής ε, Καθάρισης Τραπεζών, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και από όσο ξέρω μόνο άντρες είναι υποψήφοι ε, για αυτά τα αξιώματα. Ίσως θα πρέπει να θυμίσουμε στο Συμβούλιο ότι καλό είναι να μας προσιάζουν λίστες υποψηφίων που να έχει ίδιο αριθμό ανδρών και γυναικών να προσπαθήσουμε να έχουμε μια πιο σφαιρική εικόνα, διότι ε, προχωράμε έτσι τμηματικά και τελικά περισσότεροι άνδρες είναι αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν αυτά τα αξιώματα. Για την επόμενη έκθεση όμως, γιατί με βέβαια θα υπάρξει η επόμενη έκθεση, καλό θα είναι η κυρία μου να μας προτείνετε συγκεκριμένες, συγκεκριμένες προτάσεις τι σημαίνει ένα προπολογισμό που αναλαμβάνει υπόψη την ισότητα των δύο φύλων. Θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρό σας, ε, ο οποίος ε, θα σας μιλήσει για τα επίγοντα μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στα πλαίσια του Brexit. Ως εισηγητής ε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ο Επίτροπος Έτιγκερ παρουσίασε την πρόταση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συνεδρίαση της 7 Η Φεβρουαρίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε γραπτός απαντήσει σε ερωτήματα του Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Προπολογισμού. Θα ήθελα να εξηγήσω ότι εγώ είμαι υπέρ του να υποστηρίξουμε του σχεδιοκανονισμό. Είναι προ συμφέρον όλων να αποφύγουμε μια απότομη ε, λήξη η διακοπή τη εφαρμογή των προγραμμάτων τη Ένωση. Αυτό είναι προ συμφέρον και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και των δικαιούχων που βρίσκονται στη χώρα αυτή, των δικαιούχων των προγραμμάτων αυτών. Ε, θα ήθελα βεβαίω το Βρετανικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει το, τη συμφωνία εξόδου έτσι ώστε να μην έχει λόγο ύπαρξη αυτό το σχέδιο κανονισμού. Θα ενημερωθούμε επ' αυτού εντός των επόμενων ημερών. Αυτή όμως η επιθυμία δεν ξέρουμε αν θα, θα γίνει πραγματικότητα και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Σε ό,τι αφορά τώρα το χρονοδιάγραμμα. Ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει μόνο εφόσον αναλάβει επισήμως το θέμα το, το Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο. Κάτι που δεν θα συμβεί αν το, Ευρωπαϊκό, το, το Βρετανικό Κοινοβούλιο εγκρίνει το, στην συμφωνία. Ε, μιας και η διαδικασία θα σταματήσει. Αν όμως το Βρετανικό Κοινοβούλιο ζητήσει μια μικρή παράταση σε σχέση με την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 50 της συνθήκης, μια μικρή παράταση ή μια μεγαλύτερη παράταση, αν γίνει αποδεκτή, αυτό το αίτημα παράτασης, τότε Μόλις τον Ιούνιο θα ενημερωθούμε, θα, μάλλον θα αναλάβουμε το ζήτημα. Η επόμενη λοιπόν ε, ολομέλεια θα τον αναλάβει το επόμενο κοινοβούλιο. Θα δώσω τώρα το λόγο στους ε, συντονιστές των πολιτικών ομάδων, δύο λεπτά ο καθένας, εφόσον το επιθυμείτε και οποιοδήποτε άλλος βεβαίως στη συνέχεια θέλει το λόγο για ένα λεπτό. κύριος Φερνάντες θα μας πει την άποψή του. Επιφυλάσσεται η κυρία Θάουαλ. Νομίζω ο κύριος Φερνάντες θα συμφωνήσει μαζί μου. Μάλλον συμφωνούμε με την, ε, με την πρόταση. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, λέει ο Πρόεδρος. Ε, το Συμβούλιο δεν μας είπε ποια είναι η πρότασή του. Ο εισηγητής σας ε, βεβαίως ε, είναι καλοπροαίρετος. Ε, θέλει να κάνει ό,τι είναι χρησιμότερο και ωφελημότερο για τα συμφέροντα της Ένωσης. Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο. η υποστήριξή σας και η εμπιστοσύνη προς τον εισηγητή πραγματικά χαροποιούν τον εισηγητή. Ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και με την Ευρωζώνη. Θα κλείσω ενημερώνοντάς σας ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι Μαρτίου, 4 το απόγευμα. Όσοι θέλουν το Κοινοβούλιο να μην συμφωνήσει, να μην συνενέσει, δεν χρειάζεται να υποβάλουν τροπολογίες αρκεί να ψηφίσετε κατά του σχέδιου ψηφίσματος. Τώρα θα δούμε τα επόμενα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Και θα δώσω το λόγο τον Ντανιέλε Βιώτη πρώτα, το εισηγητή του προπολογισμού 2019, και στην Μόνικα Χολμάιερ, που είναι εισηγήτρια για το προπολογισμό του 2020. Κύριε Βιώτη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Στη διάρκεια της ε, δημοσιονομική διαδικασίας του 2019 υποβλήθηκαν 344 τροπολογίε για την εισαγωγή ε, πιλωτικών και προπαρασκευαστικών ε, project. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για τους ευρωβουλευτές. Τα πιλωτικά project και οι προπαρασκευαστικές δράσεις επιτρέπουν, θέλω να το θυμίσω, ε, την, επιτρέπουν τον πειραματισμό σε νέε πολιτικέ που θα μπορούσαν να μετατραπούν σε προγράμματα και ευρωπαϊκέ δραστηριότητε για να ανταποκριθούμε σε νέε προκλήσει. Το project του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για το 2018 περιλάμβανε 75 ε, πιλωτικά project και προπαρασκευαστικές δράσεις. Μια συμβιβαστική στηρίχθηκε στην πολιτική στήριξη το project από το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και στην αρχική του εκτίμηση από πλευράς τη Ευρω... της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, συνολικά το 2019, για το 2019 έχουν προβλεφθεί 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι αντίστοιχο στο ανώτατο όριο που ορίζεται από τον δημοσιονομικό κανονισμό. Όσον αφορά τα προπαρασκευαστικέ δράσεις έχουν προβλεφθεί 74,93 εκατομμύρια ευρώ για τις δράσεις που προτείνει το Κοινοβούλιο και ε, σε αυτά προστίθεται 25 εκατομμύρια για την έρευνα και για την, για την άμυνα που ήδη έχει ξεκινήσει και έτσι φτάνουμε περίπου στα 100 εκατομμύρια που προβλέπει ο δημοσιονομικός κανονισμός. Στην υλοποίηση των project των προπαρασκευαστικών και των πιλωτικών που έχουν εγκριθεί το 2019, η Κομισιόν μας ενημερώνει ωστόσο ότι τα δύο πιλωτικά project καλύπτονται από τη νομική βάση. Το ένα είναι το Carbon Firm και το άλλο είναι Investing in Sustainable Peace και Community Rebuilding στην περιοχή Κάουκα της Κολομβίας και δύο άλλα project είναι το Space Traffic Management ε, και το άλλο είναι η Consumer Organization στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, τώρα ξέρουμε τι γίνεται με τα πιλωτικά του 19. Η Μόνικα Χολμάγερ για τον προπολογισμό 2020. Αγαπητέ πρόεδρε, συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε το έγγραφο εργασία σε ό,τι αφορά τα παιδικά προγράμματα και σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικέ δράσει για το διαδικασία 2020. Έχουμε δύο προθεσμίε για τι προτάσει PPA και για πρώτη αξιολόγηση. Πρώτο γύρος 8 Απριλίου, το μεσημέρι στι 12, δεύτερο γύρο, 11 Ιουλίου το μεσημέρι. Γιατί αυτό ο δεύτερο γύρο, γιατί αυτό έχει να κάνει με τη θητεία από τον Ιούλιο και μετά θα έχουμε του νέου συναδέλφου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν και αυτή την ευκαιρία, εφόσον το επίθυμουν, να κάνουν κάποια πρόταση. Ακόμα και αν δεν συμβεί κάτι στην πράξη, πρέπει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα μέλη λοιπόν του Μερεντικού ε, Κοινοβουλίου στην 8 θητεία θα μπορέσουν να συμμετέχουν μόνο στην πρώτη, στον πρώτο γύρο και μόνο τα εκλεκθέντα μέλη στο δεύτερο γύρο. Δεν θα ήταν καλό τα παλιά μέλη τα οποία θα επανεκλεγούν να έρθουν και να προσπαθήσουν να ξαναπεράσουν αυτά τα οποία έχουν συζητήσει ήδη στον πρώτο γύρο. Αυτό θα οδηγούσε σε, σε κακή ε, αξιολόγηση. Καλό θα ήταν λοιπόν επίσης να μην προταθούν τα θέματα αυτά με καινούργιο όνομα, αλλά συμφωνήσουμε, γιατί ε, το δεν θα τα προλάβουμε κιόλα. Είναι τόσο πολλά αυτά τα πολιτικά προγράμματα. Άρα όλοι όσοι είναι στο Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να έχουν την 8η Απριλίου ε, στο κεφάλι τους για το κατά πόσο θέλουν να προτείνουν κάποιε παρασκευαστικέ αρχέ δράσει και κάποια πλωτικά προγράμματα. σε ό,τι αφορά τα σχέδια τροποποίηση του προπολογισμού, μόνο τα πλήρη μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής ε, Προπολογισμού μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις αυτές. Ε. Τα άλλα μέλη μπορούν να υποβάλουν ε, τέτοιες προτάσεις εφόσον είναι ένας από τους συγγραφείς της πρότασης μόνιμο μέλος. Γιατί από τις εκθέσεις του Ντανιέλα και του Ζικ πρέπει να πούμε ότι είχαμε κάποιες εμπειρίες, ότι τελικά είχαμε κάποιες ε, α, τροπολογίες οι οποίες δεν είχαν να κάνουν τίποτα ουσιαστικά με το αντικείμενό μας ως Επιτροπή Προϋπολογισμού και γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να το λάβουμε αυτό υπόψη. Και έτσι συμφωνήσαμε επ' αυτού. Οι ειδικέ επιτροπές αν δεν θα πρέπει να ορίσουν ανώτατο όριο Κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται μία φορά και μόνο και οι προτάσεις, ε, αν είναι δυνατόν, θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά ή στα γερμανικά γαλλικά. Έτσι θα απλοποιούσαμε την ε, αντίδραση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σε εγκαίρο τουλάχιστον. Γιατί δάλλω έχουμε και τις μεταφράσεις και δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Δεν θέλουμε να σημαίνει αυτό περιορισμό των γλωσσών, ούτε σημαίνει αυτό ότι δεν θέλουμε συστηματικά να υπάρχουν άλλες γλώσσες. Είναι χρονικός ο περιορισμός μόνος. Οι προτάσεις θα διατεθούν μέσω του έντυπου στο e-committee. Είναι τυποποιημένο και σας παρακαλώ να το χρησιμοποιήσετε. Τα τελευταία χρόνια είχαμε διάφορους που από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ε, έβαζαν α ή β άμα ως προτεραιότητα, αν φυσικά υπάρχει εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εκτίμησε σωστά την προτεραιότητα από πλευρά του Κοινοβουλίου, μπορούμε να υποβάλουμε ένσταση. Ύστερα, σε θέματα ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας, εκπαίδευσης, θέματα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αυτά είναι θέματα προτεραιότητας και σίγουρα θα αναδεχθούν ως θέματα προτεραιότητας εκ νέου και σε ό,τι αφορά και την πολιτική γειτονία, σε αυτόν αναλογεί και μάλλον αντιστοιχεί και με τις κατευθυντήριες γραμμές μας. Όλες οι προτάσεις που πρέπει να υποβληθούν τον Απρίλιο και τον Ιούλιο θα υποβληθούν και για τον Σεπτέμβριο ως πρόταση τροποποίησης του τροπολογισμού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό λοιπόν, Πρόεδρε, για να σας επενθυμίσω τα γενικά και τα βασικά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. αυτή και αν έχετε κάποια ερώτηση, φυσικά είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άρα, το μήνυμα προς τους ε, βουλευτές ε, της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού είναι σαφές. 8 Απριλίου είναι η προθεσμία και τον Ιούλιο δεν έχουμε ουσιαστικά μια μεταξυστική περίοδο. Είναι για τους μελλοντικού βουλευτές αυτή η δεύτερη προθεσμία. Ο σκιώτης συζητής τώρα έχει το λόγο. Είναι μάλλον οι σκιώδες που θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν βλέπω κανένα να ζητάει το λόγο. Άλλοι συνάδελφοι. Αν θέλει κανείς να πάρει το λόγο, να το ζητήσει τώρα. Έτσι φαίνεται. Ο κύριος Βιώτη και η κυρία Χολμαϊερ, οι εισηγητές ήταν τόσο σαφείς που δεν υπάρχει καμία περαιτέρω ερώτηση. Ίσως ο κύριος Ουρέλ θα ήθελε να πάρει το λόγο να μας παρουσιάσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω τον κύριο Βιώτη και την κυρία Χολμάιερ για την παρουσίασή τους. Ε, εμείς συμφωνούμε απολύτως η ενδιάμεση έκθεση της Κομισιόν που παρουσίασε εν συντομία ο Βιώτη δείχνει ότι η διαδικασία που έχουμε θεσπίσει λειτουργεί καλά. Η συντηρητική πλειοψηφία των πλειοτικών προγραμμάτων και των προπαρασκευαστικών δράσεων που επελέγησαν και ψηφίστηκαν εφαρμόζονται όπως προβλεπόταν και νομίζω ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό έγινε χάρη στο προπαρασκευαστικό έργο την αξιολόγηση της Κομισιόν και τις εργασίες του Γενικού Εισηγητή που εξετάζει πολύ προσεκτικά αυτήν την αξιολόγηση. Αυτό νομίζω οδηγεί σε μια πολύ καλή εφαρμογή σε πολύ καλά αποτελέσματα εφαρμογή. Τώρα αυτό το έτος έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι θα έχουμε το δεύτερο γύρο αξιολογήσεων που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το καλοκαίρι σας διαβεβαιώ ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να το κάνουμε αυτό όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι θα είναι καλοκαίρι ε, και θα δυσκολευτούμε να βρούμε όλους τους συναδέλφους ε, στα γραφεία τους. Πάντως ε, η Κομισιόν θα συνεργαστεί στο μέτρο του δυνατού για να σου παρουσιάσει την αξιολόγηση του συντομότερο. Και βέβαια όσο πιο γρήγορα λάβουμε τις νέες προτάσεις, το δεύτερο γύρο προτάσεων του Κοινοβουλίου, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε να τα μελετήσουμε. Τελειώνοντα, να πω ότι δεν έχω καμία απολύτω αμφιβολία ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την κυρία Χολμάιερ, όπω και με τον κύριο Βιώτη πέρυσι. Και περιμένουμε με μονησία αυτή τη συνεργασία. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ιουρέλ. Τελειώσαμε, λοιπόν. Ολοκληρώσαμε Ε, τα, τα σημεία πέντε ψηφοφορία διακόπτουμε έως τις 12 διότι στις 12 είναι προγραμματισμένη η ψηφοφορία διακόπτουμε λοιπόν Chers collègues, la séance est reprise. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία των συμβαστικών προτάσεων και των τροπολογιών για το σχέδιο έκθεσης κατακτήριων γραμμών της κυρίας Χολμάιερ, της Γενικής Εισηγήτριας για τον προπολογισμό 2020. Θα κάνουμε πρώτα μια δοκιμή βάλτε τις κάρτες μέσα στα μηχανήματα. Άρχιτη ψηφοφορία. Non. Ça y est, vous êtes prêts Είστε έτοιμοι. Άρχιτη ψηφοφορία. L'un d'entre vous n'a pas voté. Bon, bah, le scrutin est clos. Hein. Πέρας ψηφοφορίας. Amendement de compromis numéro 1, qui est pour. Συμβασμός 1, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβασμός 2, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβασμό 3, υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνδεσμός 27. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο μέρος της τροπολογίας 27 παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Μάλιστα. 18 υπέρ, ε, μάλλον 14 ε, υπέρ, 18 κατά απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασ... Ε, όχι, τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 19-11. Συμβασμός 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συ... Ε, τροπολογία 49. Προ... Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 71. Με ξεχωριστή ψηφοφορία, πρώτο μέρος. Α, συγγνώμη. Το πρώτο μέρος έχει καλυφθεί. Δεύτερο μέρος, υπέρ. Κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται τροπολογία 73 σε δύο σκέλη για το δεύτερο μέρος του 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβασμός 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 79 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ για το πρώτο μέρος του 79. Πέρας ψηφοφορίας. Μισή-μισή. Που σημαίνει ότι απορρίπτεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 87. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 17-15. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 99 τροπολογία. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πρώτο μέρος του 99. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται 17-16 Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο μέρος του, 10, του 99, συγγνώμη, τροπολογής 99. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 17-16. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107. Α, όχι, καταπίπτει. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβασμός 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε για την τροπολογία 2 άρχιτη ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 17-16 τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 3 Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 19-14. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επί του συνόλου του κειμένου τώρα. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 7 κατά 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον Γενικό Εισηγητή. La parole est maintenant au rapporteur général. Και τώρα το λόγο έχει ο Γενικό Συγητή του Προλογισμού του 2019, κ. Βιάτη, για κάποιε μεταβιβάσει, κάποια βάσματα στο του 2019. λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε τρία αιτήματα για μεταφορές 80 εκατομμύρια υποχρεώσεις από την ε, αποθεματικό ε, πληρωμές ε, προς την Τουρκία ώστε να εξασφαλιστεί η επισητιστική βοήθεια για την Ιεμένη όπου εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε κατάσταση λοιμού. Μάλιστα η κατάσταση θα επιδεινωθεί από ό,τι προβλέπετε, γι' αυτό προτείνω την υπερψήφιση. Δεύτερο αίτημα 3 του 2019 είναι 30 εκατομμύρια ευρώ και 40 ε, ε, εκατομμύρια από την ε, συμφωνία για την, από τη γραμμή μάλλον για την Τουρκία είναι για να ε, βοηθηθούν πάλι οι κατάσταση των προσφύγων που επιδεινώνεται επικίνδυνα. 24 εκατομμύρια είναι οι τέσσερα για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στο νότιο Σουδάν, η πιστιστική βοήθεια δηλαδή, υπέρ των προσφύγων στο Σουδάν και στην Αιθιοπία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Σίτα. Και τώρα θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική κλίση και ίσως ο κύριος Χουρέλ να μπορούσε να μας δώσει κάποιες περαιτέρω διευκρινήσεις. Όχι, Πρόεδρε. Ο εισηγητής ήταν σαφής και θέλω να τον ευχαριστήσω για την σύσταση υπερψήφισης των τριών προτάσεων που πιστεύω θα δώσουν ενισχύσεις πέρα από αυτά που είχαν ήδη ε, προβλεφθεί στον ψηφισμένο προπολογισμό για αυτές τις τρεις μεγάλες κρίσεις. Ευχαριστώ. Θα περάσουμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία με ηλεκτρονική κλίση. Για το 02 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ και μια αποχή. Το 03 επίσης άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ και μια αποχή. Για το 04 άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ, μία αποχή. Κύριε Γενική Εισηγητά, έχουμε επίση ε, ε, τροποποίησεις, αλλαγές ε, στο πίνακα της Επιτροπής. Ναι, η Κομισιόν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το άρθρο 53 του Δημοσιονομικού Κανονισμού για να μετατρέψει 130 θέσεις ΑΣΤ μόνιμες σε SC. Ε, για το οργανόγραμμα της ε, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για έμεσες δράσεις. Ε, σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρήση του προεπισοπικού SSC θα επιτρέψει ε, μια εξοικονόμηση και επιτάχυνση το 2019. Αυτά γίνονται επί τη βάση του άρθρου 53 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, αφορά αντί 16, 15 και 14 και τουλάχιστον το 10% των επιτρεπόμενων θέσεων ε, που προβλέπονται από το οργανόγραμμα. Ο όγκος ε, δε των αποδοχών ε, σε σχέση με ολόκληρο το χρόνο είναι μειωμένο και το όριο δεν ξεπερνιέται. Ωστόσο, ε, μπορούμε να διερωτηθούμε γιατί η Κομισιόν φτάνει τώρα με μια τόσο σημαντική αλλαγή και δεν ήταν δυνατόν να γίνει μέσα στο διορθωτικό προϋπολογισμό που συμφωνήσαμε πέρσι στο δεύτερο, ή στο δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, ευχαριστώ. Κύριε Ιουρέλ, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση του Γενικού Εισηγητή. Γιατί τόσο σημαντικές αλλαγές λίγες εβδομάδες μετά την έγκριση ε, του προϋπολογισμού. Uh, yes, thank you, Chairman, and thank you to the... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Κατανοώ την ερώτησή του. Είναι θέμα χρονικής συγκρίας. και αντιληφθήκαμε την ε, ανάγκαιότητα της αλλαγής αυτής μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και ως εκ τούτου συνεχίσαμε τη διαδικασία όπως προβλέπεται από το άρθρο 53 του οικονομικού κανονισμού. Σημειώνω προφανώς στο σχόλιο του εισηγητή. Ότι προφανώς το μέλλον θα ήταν πιο σωστό να γίνεται εκ των προτέρων η αλλαγή αυτή. Ευχαριστώ. Μάλιστα, συναδελφοί, είναι τελευταία φορά το καταγράφουμε αυτό ιστορικά ότι δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, μήπω θέλει κάποιο να πάρει το λόγο, κανεί. Μάλιστα. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρώ ότι εγκρίνεται αυτή η τροποποίηση. Ο κύριο Ρούμπιχ δεν έχει να κάνει κάποια πρόταση. Όχι κάτι παραπάνω από ότι σε σχέση με την πολιτική την Κυριακή και άρα ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Και τώρα θα συνεδριάσουμε και κλεισμένο το Να καλέσω όλους όσοι δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στη συνεδρία κλεισμένο το θυρών να εξέλθουν τις αιθούσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και σας αυτό καλό Σαββατοκύριακο.